Uh, και κύριοι, λέω να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας συνεδρίαση. Πρώτα μερικές ανακοινώσεις. Υπάρχει αναμετάδοση και όσους παρακολουθούν στο ίντερνετ τους καλωσορίζω και αυτούς και τους ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε λιγάκι. Είμαστε από τις επιτροπές με τις περισσότερες αναμεταδόσεις. Πράγμα που δείχνει πόσο τεράστιο ενδιαφέρον σημειώνεται για τη δουλειά μας. Θα ήθελα να δείτε και τα έγγραφα τα σχετικά για τη δουλειά μας γενικότερα παραδείγματος χάρη. Πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα δηλαδή έγινε μια ανακοίνωση για την αγορά ηλεκτρονικών ειδών από τους καταναλωτές και τις καταναλώστριες μέσω ίντερνετ. Μπορείτε να τα βρείτε και ηλεκτρονικά, να σας στείλουμε δηλαδή ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο του φυλαδίου μας. Ήπι Παύλα Ήμκο Παύλα Ευρωπάρλ, Παύλα ΕΟΥ, σε όποιον ενδιαφέρεται. Ίσως μερικοί να το, μπορούν να το λαμβάνουν και αυτόματα, αν βέβαια τα καταφέρει το κοινοβούλιο να οργανωθεί, λοιπόν, να αρχίσουμε ένα δίκτυο, δηλαδή οι φίλοι της ΣΥΜΚΟ και οι φίλες. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δέχεστε την ημερήσια διάταξη επισήμω, υπάρχει μια αλλαγή στη σειρά. Ένας από τους εμπειρογνώμονες δυσκολεύεται να προσέλθει. Αναμένουμε ότι σε καμιά ώρα θα καταφτάσει. Είπαμε λοιπόν να αλλάξουμε τη σειρά και να συζητήσουμε πρώτα το δεύτερο θέμα της κυρίας Στάιλερ για τις δομικές κατασκευές. Και θα μας μιλήσει βέβαια και η Κομισιόν. Με αυτή την αλλαγή μπορείτε να εγκρίνετε την μισή διάταξη άψογα. Ευχαριστώ. Και στο τέλος σας καλώ όλους και όλες σε ένα κοκτέιλ το σαλόνι των βουλευτών στις 6.30 για να γιορτάσουμε την πέμπτη επέτειο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταναλωτών και Καταναλωτριών. Τι είναι αυτό. Α, υπάρχει εδώ αυτό το φυλάδιο για την πέμπτη αυτή επέτειο. τα Χαλεταστόρη που είναι της Γενικής Διεύθυνσης Σάνκο και εγώ θα είμαστε οι συνδετημόνες ή θα σας καλέσουμε μάλλον, θα είμαστε οι αμφιτρίωνες μάλλον. Σας καλωσορίζω λοιπόν τώρα στη δεύτερη ανάγνωση για την πρόταση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Η κυρία Στάιλερ μας έχει γράψει ένα σχέδιο σύστασης που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες και θα δούμε τώρα που βρίσκεται η εξέταση. Δυστυχώ, ο κύριος Μάγερ δεν έχει έρθει, δεν ξέρω αν συνεννοήθηκε με κανέναν. Ο κύριος Μπουζόη θα μιλήσει για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Μακλάκ θα ερχόταν αλλά ίσως έρθει αργότερα, αλλιώς η κυρία Σαλβίνη. Ο κύριος Ζακ Φαρτές από το Συμβούλιο Έρχεται, καλά έρχεται. Και ο κύριος Λέος Αγκούρες. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πώς θα έχει η διαδικασία. Η προθεσμία κατάθεση των κολογιών λήγει στις 19 Οκτωβρίου και ελπίζουμε σε έκτακτη συνεδρίαση 8 Νοεμβρίου να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τη σύσταση της κυρίας Τάιλερ και έτσι να πάμε στην Ολομέλεια του, 2000, του Ιανουαρίου 2011 για να ολοκληρωθεί έτσι η δεύτερη ανάγνωση. Μάλιστα. Και τώρα το λόγο έχει η συγγήτριά μας κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε και εσάς και τους κοιόδης καθώς και όλους όσους ήρθαν στην ακρόασή μας την περασμένη εβδομάδα για, τα δομ... για τις δομικές κατασκευές. Ήταν πολύ χρήσιμη υπήρξε. Έντεκα ομιλητές και ομιλήτριες πήραν το λόγο. Και οι συνάδελφοι που ήρθαν άκουγαν πολύ προσεκτικά, το παρατήρησα. Θα ήθελα λοιπόν για να μην επαναλάβω αυτά που είπα τότε, οπότε και είχα δηλώσει ότι οι καλοί φράχτες κάνουν τους καλούς γείτονες. Θα περιοριστώ μόνο στο θέμα των δηλώσεων αποπεράτωσης, το θέμα των ε, τοξικών υλικών που δεν είχε συμπεριληφθεί αρχικά στην κοινή θέση, το θέμα της διαφάνειας και το θέμα της επαφής με ορισμένα συγκεκριμένα υλικά. Και γενικότερα το θέμα υγείας, αλλά και επικοινωνίας και της ανάγκης να υπάρχει συνοχή στα συμβόλαια και υπόλοιπα έγγραφα. Έχει τεθεί και το θέμα της χρηματοδότηση e ορισμένων υλικών έχουν ζητηθεί εξαιρέσεις, θα τις εξετάσουμε και αυτές. Τις επιτήρησης, τι πρέπει να δηλώνεται και τι δεν πρέπει η διαφορά μεταξύ εργολάβων και κατασκευαστών, η ασφάλεια μερικών προϊόντων. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι έχουν τη μετάφραση στη γλώσσα τους. Σήμερα δυστυχώς δεν μπορώ να παραμείνω στο κοκτέιλ στις 6.30 γιατί έχουμε συνάντηση σκιωδών με την Κομισιόν για να δούμε ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες και αν υπάρχει καμία συνένεση. Δεν έχω δυστυχώς τίποτε άλλο να προσθέσω. Μόνο το ότι έγιναν οι μεταφράσεις. Απλώς σας θυμίζω ότι η διορία κατάσταση τροπολογιών λήγει στις 19 Οκτωβρίου και θα υπάρξει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 8 Νοεμβρίου. Σας Παρακαλώ λοιπόν αν ενδιαφέρεστε για δομικά υλικά να καταθέσετε γέρο στις τροπολογίες σας ε, γιατί θα θέλαμε να συζητήσουμε ισκιώδης με την Προεδρία έγκαιρα για να υπάρξει επαναλαμβάνω για όσους δεν το κατάλαβαν κάποια συνένεση και τώρα με χαρά να ακούσω αν έχετε κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Στάιλερ. Σας ευχαριστώ θερμά καταρχήν για τη διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης που όπως είπατε ήταν πολύ ενημερωτική και περιεκτική. Γιατί και εσείς και οι σκιοδησηγητές ε, επιτελείτε πολύ σημαντικό έργο. Θα περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος Βάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο γιατί ο κύριος καθηγητής Μάιερ, ο σκιώδη εισηγητής μας δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα έρθει το βράδυ. Θα ήθελα να ευχαριστήσει τον, ε, την εισηγήτρια για την ε, επικοτομητική συνεργασία και να πω ότι εξ ονόματο του ΕΛΚ η διάκριση των μικροεπιχειρήσεων δεν ε, είναι ε, η κατάλληλη απαραίτητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τον όγκο των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να είναι πιο κατάλληλη η απλοποίηση της σήμανσης CE. Αλλά το να διατίθενται τέτοια προϊόντα στην αγορά που θα μπορούσαν να αποπούν επικίνδυνα, αυτό νομίζω ότι δεν θα αποβεί οι καταναλωτοί, αλλά ο καθηγητής Μάιερ, όπως σας είπα, είναι αισιόδοξο ότι θα βρει λύση με την συγκεντρία. Ευχαριστώ. Ah, ο κύριος Μπουζόη. Σας ευχαριστώ. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι από τους πιο σημαντικούς της οικονομίας και η η υιοθέτηση του νέου κανονισμού για τα δομικά προϊόντα θα άρει τους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την κυρία Τάιλερ, γιατί πραγματικά εργάστηκε άοκνα και ιδιαίτερα κατά τις θερινές διακοπές. Θα συμφωνήσω με την προσέγγιση της συγκεκριάς μας και στη συνάντηση με τους σκιώδεις ηγητές το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα την υποστηρίξω γιατί προσπαθεί να βρει μια σωστή ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των δομικών προϊόντων αλλά και της ανάγκης να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εργάζονται στον ε, κατασκευαστικό κλάδο. Είμαι υπέρ αυτών των contact points για τα προϊόντα και θα ε, πρέπει να τα εφοδιάσουμε το κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και οι διανομή τέτοιων δομικών προϊόντων θα πρέπει να ε, ενθαρρυνθούν να ζητούν πληροφορίες από αυτά τα σημεία επαφής, τα contact points και άλλο πολύ σημαντικό πράγμα είναι, όπως επισήμανε η κυρία Τάιλερ, είναι της ανεξαρτησίας αυτών των contact points από, το, από άλλα σώματα και από τις διαδικασίες για τη χορήγηση του σήματος ε, σε ε. Επίσης ε, θα πρέπει να αναλαμβάνονται δράσεις και να επιβάλλονται κυρώσεις κατά των κατασκευαστών που χρησιμοποιούν ε, εσφαλμένα το, τη σήμανση σε «ε». Το θέμα της δήλωσης απόδοσης, ε, Declaration of Performance, θα πρέπει να αποσαφινιστεί ότι ο κατασκευαστής είναι αυτός που καταρτίζει τη δήλωση απόδοσης, γιατί δεν προκύπτει αυτό με σαφήνεια από τον κανονισμό του Συμβουλίου. Θα πρέπει το προϊόν αυτό να καλύπτεται από, τις, από τα πρότυπα για τα οποία έχει εκδοθεί η ευρωπαϊκή αξιολόγηση. Συμφωνώ λοιπόν με την προσέγγιση κυρία κυρία Στάιλερ, γιατί χάρη στην έκθεσή της θα αποσαφινιστεί η κατάσταση και θα αρθούν οι φραγμοί στην εσωτερική αγορά δομικών προϊόντων. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπουσόη. Η κυρία Ρούλε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Στάιλερ και όπως είπατε ήταν πραγματικά πολύ καλή δουλειά της και έβαλε στο κείμενο αυτά που θέλαμε από την πρώτη ανάγνωση και δεν είχε αποδεχτεί το Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω όμως και το Συμβούλιο γιατί στην πρώτη ανάγνωση ε, ενέκρινε πολλά στοιχεία τα οποία θέλουμε να τα κρατήσουμε και στην δεύτερη ανάγνωση. Μόνο λεπτομέρειες έχω να σχολιάσω και θα υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του μνημείου και κατά πόσο προέρχεται από τη δεκαετία του 50, αν είναι παραδοσιακό κτίριο. Για μένα υπάρχουν κάποιες μικρές έτσι, λεπτομέρειες και αυτό που είπε και ο κ. Σφάμπ για τις μικροεπιχειρήσεις. Να προσέξουμε το εξής, γιατί οι πιο πολλές μικροεπιχειρήσεις χρειάζονται τις κατάλληλες πληροφορίες για να αναλαμβάνουν και το σχετικό ρίσκο σε ό,τι αφορά την, ε, τα προϊόντα αυτά. Άρα, θέλουμε μικροεπιχειρήσεις από πλευράς των κατασκευών, αλλά και μικροεπιχειρήσεις από πλευράς των προϊόντων. Θα υποβάλω λοιπόν σχετικά κάποιες τροπολογίες. Uh, uh, Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια εκ μέρους κυρίας Μακλάρκιν. Καταρχήν, και εμείς υποστηρίζουμε τις βελτιώσεις που επέφερε το Συμβούλιο στην πρόταση, όπως είπε η κυρία Ρούλε. Και μας επόμεναν κάποιες κρίσιμες λεπτομέρειες. Θα πρέπει πάντως να εμείνουμε στις βελτιώσεις και κυρίως ε, να πλουστεύσουμε το γραφειοκρατικό άχθος ε, για το κατασκευαστικό κλάδο, ιδιαίτερα με την κατάργηση της υποχρέωσης πολλαπλών δηλώσεων. Είναι πολύ θετική αυτή η βελτίωση και μην ξεχνάτε ότι πολλές είναι πολλοί άριθμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο. Η κυρία Ρούλε αναφέρθηκε στους ε, ειδικευμένου που ασχολούνται με την αναπαλαίωση ιστορικών μνημείων νικτηρίων και εκεί ενδιαφέρει όχι μόνο η ποιότητα και η χρήση των υλικών αλλά και η ελάφρυνση της υπερβολικής γραφειοκρατίας. Επίσης το θέμα της ελεύθερη διακίνηση. Όλα αυτά είναι σημαντικοί στόχοι, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Οι, τροπο, οι τροπολογίες της σε αυτή την κατεύθυνση ακολουθούν και θα πρέπει να μείνουμε σε αυτές τις βελτιώσεις, χωρίς όμως να επιβαρύνουμε το θέμα της ασφάλειας ή να το διακυβεύουμε. Η κυρία Στάιλερ ίσως αργότερα σχολιάσει το επίμαχο ζήτημα των επικίνδυνων ουσιών. Θα πρέπει οι σχετικές διατάξεις να μην επαναλαμβάνουν ε, τις διατάξεις του Ρίτσι, να μην επιβάλλουν ε, υπερβολικό άχθος για ορισμένα προϊόντα και για κατασκευαστές που ήδη έχουν δηλώσεις ε, επικίνδυνων ουσιών σε ορισμένα από τα προϊόντα που παράγουν. Ίσως ήθελα να το σχολιάσει η κυρία Στάιλερ, γιατί προς το παρόν διαφωνούμε με το Συμβούλιο, αλλά ελπίζω να καταλήξουμε συμβαστική λύση μαζί του για το θέμα των επικίνδυνων ουσιών. Αυτά έχει να πει η κυρία Μακλάρκιν και και γήτρια. Θα δώσω τώρα, αν δεν έχει αντίρρηση η κυρία Στάιλερ, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία, στην Βελική Προεδρία. Πρώτα θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Λέο Αγκουέγες, για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, αν εδώ ε, θα καταφθάσει ένα πάσα στιγμή ο κ. Πέτρασον το ελπίζουμε. Στο μεταξύ όμως θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω κι εγώ τα συγχαρητήριά μου προς την εισηγήτρια για την πολύ αξιόλογη της έκθεση. Είναι τόσο αξιόλογη και καταπληκτική που σχεδόν συμφωνούμε στα πάντα με την εισηγήτρια. Γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στις συστάσεις σας συμβάλλουν γενικώ στη βελτίωση και εμπλουτισμό της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε να δεχτούμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες σας. Ναι μεν, αλλά, γιατί υπάρχει και ένα αλλά. Το γνωρίζετε άλλωστε. Όπως το ανέφερε και ο Πρόεδρος, το αλλά αφορά τη σχετική τροπολογία για τις επικίνδυνες ουσίες. Hazardous substances. Είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας η ισχύουσα νομοθεσία που είναι και πολύ δυναμική, δηλαδή εξελίσσεται, δεν είναι στατική, εξελίσσεται μέρα με τη μέρα και εν ανάγκη μπορεί να συμπεριλάβει και νέες τέτοιες ουσίες. Πιστεύουμε ότι είναι αρκετή αυτή η φυστάμενη νομοθεσία και είναι και η εφαρμοστέα νομοθεσία. Και αυτή θα πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς και να το οποιαδήποτε επικάλυψη. Πολλά δε μάλλον που πριν από λίγο μάθαμε ότι στη Γερμανία καταρτίστηκε μία μελέτη από μία εταιρεία συμβούλων με θέμα τις επιπτώσεις που θα είχε για τις επιχειρήσεις ε, η συμπερίληψη του νέου καταλόγου ουσιών που προτείνει η τροπολογία σας. Μόλις το πρωί φυσικά ε, κοίταξε εντάχει μια σύνοψη αυτή τη γερμανική έκθεση, από την οποία προκύπτει με σαφήνεια ότι για ορισμένε μικρομεσαίε επιχειρήσει το γραφειοκρατικό επιπλέον άκθος θα είναι δυσβάσταχτο. Και υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτηματικά που ανακύπτουν με την τροπολογία αυτή για τον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών. Τι ακριβώς απαιτείται και πώς θα πρέπει οι επιχειρήσει αυτές να χορηγούν τις σχετικές πληροφορίες. Όλα αυτά είναι κάπως ασαφή και προσδιορίστα. Ω εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς δεν μπορεί να δεχτεί την τροπολογία σας αυτή. Θα ήθελα να υποβάλω και ένα σχόλιο για ένα άλλο σημαντικό θέμα, αυτό που επισήμανε η κυρία Ρούλε, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υπόψη περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα και όχι αυτές που τα χρησιμοποιούν τα καταναλώνουν. Πάντως θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και την αντίθετη ερμηνεία. Δηλαδή, Στην πρόταση αυτή κανονισμού έχουμε τη μόνη περίπτωση όπου ο κατασκευαστής έχει την υποχρέωση να πει ότι το προϊόν που θέτει στην αγορά πληρεί τις ε, ισχύουσες διατάξεις και τις ε, προδιαγραφές. Είναι η μόνη φορά που η εταιρεία που χρησιμοποιεί το προϊόν μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα πρόβλημα γιατί γνωρίζει ότι πληρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις που πρέπει να αναφέρονται στην δήλωση απόδοσης της κατασκευάστριας μικροεπιχείρησης. Χάρη σε αυτή τη δήλωση, ξέρει ότι το η εταιρεία που χρησιμοποιεί το προϊόν ξέρει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας και ως εκ τούτου μπορεί άφοβα να το χρησιμοποιήσει. Με το άρθρο 37 και οι δύο επιχειρήσεις βγαίνουν κερδισμένε από άψη κόστους. Και η κατασκευαστική επιχείρηση που θέτει το προϊόν σε εμπορία στην αγορά, αλλά και οι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Μην ξεχνάτε ότι η διατύπωση του άρθρου 37 που προβλέπει ότι η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει ποιες προδιαγραφές πληρούνται για το προϊόν και συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις είναι τοπικές επιχειρήσεις και μπορούν κάλλιστα να εντοπίσουν τις εφαρμόσιμες απαιτήσει. Και αυτό είχε κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπέβαλε την πρόταση. Είχαμε κατά νου αυτές τις τοπικές επιχειρήσεις που συνιστούν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό δίκτυο σε συγκεκριμένες περιοχές και υποβάλλονται σε πολύ νομοθετικές διατάξεις. Μπορούν να αποδείξουν ότι το συγκεκριμένο προϊόν που θέτω σε εμπορία πληρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις. Το άρθρο 37 βέβαια τροποποιήθηκε κάπως από το Συμβούλιο και θα πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο περαιτέρω. Αυτό είπαμε και στην δημόσια ακρόαση για το Specifical Technical Documentation. Θέλουμε αυτή η διατύπωση να διαγραφεί και να αντικατασταθεί από τη διατύπωση τεκμηριώνοντας κατάλληλα τη δήλωσή τους. Δηλαδή οι μικροεπιχειρήσεις αυτές θα πρέπει με τα κατάλληλα έγγραφα, με την κατάλληλη τεκμηρίωση να δικαιολογούν να, να αποδεικνύουν ότι πληρούν την νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι το άρθρο 37 θα ευνοήσει και τι κατασκευαστικέ εταιρείε, αλλά και τις εταιρείε που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και νομίζω ότι μας ε, διευκρινίσατε κάποια χρήσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά την κοινή θέση, την οποία και ασφαλώς ε, ενθαρρύνω Δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Δεν ξέρω. Να περιμένουμε. Κυρία Στάιλερ, έχετε να σχολιάσετε μήπως από όσα ακούσατε έως τώρα. Και ίσως θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου μόλις καταφτάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις ε, παρατηρήσεις τους και για να είμαι και δίκαιη προς τον κύριο Φαντές. Νομίζω ότι φταίει το ότι αλλάξαμε τη σειρά των σημείων στην εμερήσια διάταξη. Άρα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τι έχει να πει και το Συμβούλιο όταν καταφτάσει ο εκπρόσωπος. Συνοψίζοντας, ξέρουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία χρήζουν συμβιβασμού. Ξέρουμε ότι οι επικίνδυνε ουσίε αποτελούν ένα από τα σημεία τα αμφιλεγόμενα αυτά σε ό,τι αφορά επίση και τι πολύ μικρέ επιχειρήσει τα σημεία επαφής για τα προϊόντα, η δήλωση απόδοσης. Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά συζητήσαμε και θέματα ανακυκλωσιμότητας και των στόχων των περιβαλλοντικών. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Ελπίζω η συνεδρία σήμερα το απόγευμα να αποβεί πολύ ωφέλιμη σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες ε, συμφωνίες στο μέλλον. Θα συνεργαστώ ασφαλώ και με του συναδέλφου, που έχουν να κάνουν πολλά επικοδομητικά σχόλια και χάρηκα που άκουσα τα σχόλια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την αρχική μου έκθεση. Να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Είναι σημαντικό ασφαλώ να βρεθεί συμβιβασμό. Άρα, όταν θα κατατάσσει ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου, ελπίζω να του δώσετε το λόγο, γιατί δεν φταίει αυτό, καταλαβαίνετε. Yes, well, I'm very sorry ναι, πολύ λυπάμαι για την αλλαγή των σημείων, τη σειρά των σημείων, αλλά μόλις κατέφτασε και ο καθηγητής ε, Δ. Σούλτς. Αυτός ήταν και ο λόγος που αλλάξαμε την σειρά των σημείων. Δεν ξέρω πότε θα καταφτάσει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλες πληροφορίες να μας δώσετε για τα δομικά υλικά μέχρι ότου καταφτάσει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου ή αν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να κάνει κάποιο σχόλιο. Η αν θελει κάποιο αλλος συνάδελφο Ρίλα, μήπως. Yes, I think we're here now. Yes, good. Α Ας τον αφήσουμε να βγάλει το παλτό του, να πάρει μια αναπνοή και μετά να πάρει το λόγο. Uh, um, με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν χαιρετίζουμε τον εκπρόσωπο της Προεδρίας που με τόση επιτυχία προείδρευσε των συνεδριάσεων για αυτή την οδηγία. Είχαμε αλλάξει βέβαια την σειρά γιατί είχε καθυστερήσει κάποιος προσκεκλημένος και γι' αυτό δεν μπορέσατε να παρίσταστε στην ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχει πάντως μεγάλη υποστήριξη στην Επιτροπή μας για τις βελτιώσεις που έκανε το Συμβούλιο προς την οδηγία. Και τώρα νομίζω ότι θα ήταν καλό να μας κάνετε μια ενημέρωση ως προς το πού βρίσκονται τα πράγματα στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν κοιτάξατε τις τροπολογίες της κυρίας Τάιλερ, αλλά να μας πείτε γενικότερα πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μαζί για να καταλήξει η διαδικασία εξέτασης αυτής της οδηγίας μέχρι τον Ιανουάριο. Έχετε λοιπόν το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε όλοι και όλες γιατί κάπως καθυστέρησα Δυστυχώς δεν μπόρεσα λοιπόν να ακούσω τους υπόλοιπους, αλλά αν κατάλαβα καλά αυτά που ζητήσατε, θέλετε να σας παρουσιάσω το κείμενό μας έτσι όπως έχει τροποποιηθεί τον Μάιο από το Συμβούλιο. Με βάση το κείμενο που είχε υποβάλει η Κομισιόν πριν από δύο χρόνια και τις τροπολογίες που είχε καταθέσει το Κοινοβούλιο εδώ και μήνες ξαναείδαμε, ξανααναθεωρήσαμε τη θέση μας και χρειάστηκαν συνολικά δύο χρόνια για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο αποδεκτό από όλους. Λοιπόν, ποια είναι τα κύρια σημεία που άλλαξαν. Θα προσπαθήσω να σας τα πω από μνήμης. Πρώτα πρώτα την ετικέτα ΕΕ και την δήλωση των ε, διοριών αποπεράτωσης που είναι υποχρεωτικές απόδοσης. Για τα προϊόντα που καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα τουλάχιστον ή που έχουν γίνει δεκτά τεχνικώς επανενωσιακά. Αυτό νομίζω το Κοινοβούλιο το είχε ζητήσει. Επίσης, θεωρήσαμε ότι σε μερικές περιπτώσεις έπρεπε να γίνουν δεκτές εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί από συγκεκριμένη παραγγελία για συγκεκριμένο έργο ή που τα έχει κατασκευάσει ειδικά για αυτό το έργο η εταιρεία ή αν έχουν ιστορικό χαρακτήρα ή αξία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση επειδή μερικά από αυτά είναι, χρησιμοποιούνται μία και μόνη φορά και αναπερίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν όλοι οι έλεγχοι της παραγωγής στο εργοστάσιο όπως για τα κανονικά προϊόντα. Επίσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται για συγκεκριμένα έργα θεωρήσαμε ότι όπως γίνεται γενικά στις περιπτώσεις αυτές επίσης δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη πιστοποίηση ούτε χωριστή διαδικασία που θα ήταν βαριά και δυσβάστακτη για μικρές ή ελάχιστες επιχειρήσεις. Και για τις περιπτώσεις αυτές ε, εγκρίναμε τις τρεις εξαιρέσεις που αναφέρει το άρθρο 5 για την υποχρεωτική πιστοποίηση που συμπεριλαμβάνεται στη γενικότερη δήλωση. Στην δήλωση αυτή λοιπόν θεωρήσαμε ότι, απόδοση, θεωρήσαμε ότι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της έπρεπε να είναι το εξής. Υπήρχαν πολλές λύσεις, αλλά θα μπορούσαν να είναι είτε η υποχρέωση όλα τα κύρια χαρακτηριστικά να συμφωνούν με τα πρότυπα, αυτό όμως ήταν πολύ εξαντλητικό, και για τις περισσότερες επιχειρήσεις επιβάλαμε μόνο ένα κριτήριο. Επίσης, στο άρθρο 3 προβλέπουμε η Κομισιόν να μπορεί να εφαρμόσει μία οριζόντια υποχρέωση δήλωσης Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Ξέχασα να σας πω ότι στις εξαιρεσει υπάρχουν δύο σημεία. Ένα ότι ισχύουν μόνον εάν δεν υπάρχει ανάλογη ή αντίθετη εθνική αναγκαστική υποχρέωση δήλωσης και δεύτερον η συμπερίληψη στο συγκεκριμένο έργο πρέπει να γίνεται υπό, τον έλεγχο του υπευθύνου για το έργο ή το γιαπί. Πράγμα που μειώνει σημαντικά τους πιθανούς κινδύνους που θα προέκυπταν από μία δήλωση που δεν θα ήταν συνεπής με τα πρότυπα. Αυτό ήταν το θέμα που συζητούσαμε επί δύο χρόνια. Τώρα ποια άλλα σημεία σημειώθηκαν και συζητήθηκαν ιδιαίτερα. Οι τεχνικές αξιολογήσεις, οι ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις ΕΤΑ που διαφέρουν από τις αρχικές. Αυτή τη στιγμή μια ΕΤΑ δεν μπορεί να εγκριθεί παρά μόνον εάν δεν υπάρχουν Υπάρχουν τα πρότυπα που να καλύπτουν πλήρως το προϊόν. Θα μπορούσε να υπάρχουν πρότυπα που καλύπτουν τμηματικά μερικώς το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δημοσιευθεί έτα αλλά με βάση ένα ενωσιακό κείμενο η τεχνική αξιολόγηση δηλαδή θα είναι η πρώτο, το πρώτο υποχρεωτικό έγγραφο που θα απαιτείται. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει ακριβώς αυτό γιατί έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε κατευθυντήριες γραμμές αλλά και έτα χωρίς κατευθυντήριες γραμμές, χωρίς guidelines. Πάντοτε βέβαια θα υπάρχει ένα έγγραφο τεχνικής αξιολόγησης ως πρώτο υποχρεωτικό έγγραφο. Η διαδικασία όμως συγγραφής του, σύνταξής του, αποσαφηνίστηκε λίγο-λίγο από τα άρθρα και στις προσθήκες. Πρέπει να τα ξέρουμε και τα δύο, και τα άρθρα και τις προσθήκες. Αυτά όλα βέβαια πρέπει να τα ξαναδούμε ως προς τον ακριβή τρόπο σύνταξης της τεχνικής αξιολόγησης, αλλά αυτό αναφέρουμε ότι η Κομισιόν θα το κάνει. Οι οργανισμοί που θα ευθύνονται για την σύνταξη τέτοιων εγγράφων ε, θα επιφέρουν βέβαια και κάποιο κόστος και το ε, η Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση θα έχει οριζόντιο εύρος, δεν θα καλύπτει δηλαδή ένα μόνο προϊόν, μπορεί να καλύπτει και περισσότερα. Αρχικά μπορεί να καλύπτει ένα το πρώτο τέτοιο προϊόν, στη συνέχεια όμως μπορεί να καλύπτει και άλλα. Δεν θα ήταν λοιπόν φυσικό ένας και μόνο παραγωγός να αναλάβει το κόστος της παραγωγής του κειμένου αυτού, της σύνταξης του κειμένου αυτού, και προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που να επιτρέπει την κατανομή αυτών το, αυτού του κόστους με πιο οριζόντιο τρόπο, δηλαδή να υπάρχει ας πούμε η δυνατότητα των κομισιών για την σύνταξη αυτών των τεχνικών εγγράφων. σύμφωνα και με ορισμένες τροπολογίες αλλάξαμε την αρχική θέση της Κομισιόν ως προς την τελική πιστοποίηση της τεχνικής αξιολόγησης. Το Κοινοβούλιο θέλει η δήλωση αυτή να γίνεται ηλεκτρονικά. Για μας όμως εμείς ζητήσαμε σε χαρτί Εδώ θα υπάρξουν αποκλήσεις σίγουρα. Τέλος, για να μην επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες, ένα σημαντικό σημείο απόκλησης είναι εκείνο που αφορά τις επικίνδυνες ουσίες. Στο Συμβούλιο Γίνανε πολλές συζητήσεις επί του θέματος και υπήρξε μια διαφορά μεταξύ των χωρών που ήθελαν να υπάρχει δήλωση της επικινδυνότητας ορισμένων ουσιών λίγο πολύ όπως το ζήτησε το Κοινοβούλιο και μια άλλη ομάδα χωρών που ήθελε να παραμείνει η ισχύουσα δομή από άλλες οριζόντιες νομοθεσίες και που σχετίζεται βέβαια με την ασφάλεια προϊόντων όπως το REACH ή η οδηγία για την ταξινόμηση και επιστοποίηση η οδηγία σε ΕΛΠΕ. Εκεί υπήρξε η διαφωνία στο Συμβούλιο μεταξύ των υπέρ και των κατά. Η ΔΕ ήταν, τάχθηκε υπέρ της θέσης του Κοινοβουλίου. Τελικά ζητήσαμε να συμπεριλαμβάνεται μια αιτιολογική σκέψη που να εξηγεί όλες τις, όλη την νομοθεσία που μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη δήλωση για επικίνδυνες ουσίες. Βέβαια δεν το συζητήσαμε ακόμη και γι' αυτό παραμένουμε στη θέση του Συμβουλίου να παραμείνει δηλαδή ο κατάλογος ως έχει και να μην υπάρχει υποχρεωτικός κατάλογος, υποχρεωτική δήλωση για την ύπαρξη μη ορισμένων επικίνδυνων ουσιών όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στις τροπολογίες του. Διότι οι τροπολογίες αυτές πρέπει να ξέρετε ότι τελικά ζητούσαν υποχρεωτική αναζήτηση από τους κατασκευαστές πολλών εκατοντάδων ουσιών μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν για να δουν αν είναι επικίνδυνες. Αν όμως υπάρχουν στο REACH, αν και υπάρχουν πολλές από αυτές στο REACH, παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλο το βάρος για τις μικρές ιδίως και πολύ μικρές επιχειρήσεις. γιατί φοβηθήκαμε μήπως ορισμένες επιχειρήσεις αν ήταν υποχρεωτική μια τέτοια δήλωση ζημιώνονταν υπερβολικά και γι' αυτό επιλέξαμε κάτι πολύ ελαφρύτερο και σε αυτό ακόμη βρισκόμαστε. Νομίζω ότι αν δεν απατώμε αυτά είναι όλα τα θέματα που συζητήθηκαν. Υπάρχουν και άλλα φυσικά, υπάρχουν και άλλα αλλά φοβούμε ότι για αυτά θα χρειαστούν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Α, κάτι άλλο, οι απλοποιημένες διαδικασίες. Είπαμε, και νομίζω αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο, ότι οι απλοποιημένες διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται είτε για όλες τις επιχειρήσεις είτε για τις μικροεπιχειρήσεις. 10 ανθρώπων Και για να υπάρξει αυτό προβλέφθηκαν τρία άρθρα που αναθεωρήσαμε, 36, 37 και 38. Και εκεί ζητήσαμε τη δημιουργία ενός συστήματος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μέθοδο αντικατάστασης αυτών που προβλέπουν τα πρότυπα, με την υποχρέωση όμως να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφαλείας του προϊόντος. Γιατί δεν θα ήταν λογικό να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν αυτά που προβλέπουν τα πρότυπα με οτιδήποτε, χωρίς να διασφαλίζεται η ασφάλεια. Αυτό το λέει το 37 και, και στο 2 βέβαια όπου επαναλαμβάνουμε το STD. Υπάρχει ίσως μια ασάφεια εδώ ως προς τους όρους που χρησιμοποιούνται το 36, 37 και 38 και που επαναλαμβάνεται και στον ορισμό. Γιατί αρχικά, αρχικά και για τα τρία αυτά άρθρα προβλεπόταν η λεγόμενη κατάλληλη τεκμηρίωση, όπως λέει το 2. Αλλά φάνηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο και στο 37 όπως τα υπόλοιπα σημεία και εδώ υπάρχει μια ασάφεια που πρέπει να τη λύσουμε. Και καλό θα ήταν διατηρώντας τις δυνατότητες των 36, 37 και 38 να αποσαφηνίσουμε λίγο παραπάνω πώς ακριβώς θα λειτουργεί στο μέλλον ο κανονισμός αυτός. E. Για την πιστοποίηση ή την ετικετοποίηση υπάρχει το contact point. Α, κάντε μου νόημα αν θεωρείτε ότι πρέπει να τελειώσω. Αλλά τα προϊόντα contact point είναι σύστημα που απορρέει από την οριζόντια νομοθεσία. Όπως προβλέπεται από την αμοιβαία αναγνώριση, από τον κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση. Αλλά εδώ προσθέσαμε το θέμα των εναρμονισμένων προτύπων για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ή ετικέτα. Και γι' αυτό χρειάστηκε να τροποποιήσουμε λιγάκι το σύστημα ως προς το 764 και εδώ το Κοινοβούλιο υπέβαλε μια τροπολογία όπου ζητούσε την διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας των προϊόντων contact point αυτών. η αρχή που στην οποία βασίζεται η τροπολογία αυτή δεν είναι τίποτα το περίεργο, αλλά πρέπει να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο στόχος που θέλουμε να υλοποιηθεί, ο οποίος αν δεν απατώμε είναι να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός τίμια μεταξύ των οργανισμών που χορηγούν την ετικέτα την ενωσιακή ετικέτα, η πιστοποίηση. Και θα βρούμε μια διατύπωση που να διασφαλίζει ακριβώς τον θεμητό ανταγωνισμό, διατηρώντας όμως και τη δυνατότητα για ορισμένα κράτη να προσφύγουν στα notified bodies ή σε οργανισμούς όπως τα TAB που λένε στα αγγλικά. Με συγχωρείτε που δεν το έχω μάθει γαλλικά λέει ο μιλητής, αλλά έτσι τα λέμε στο Συμβούλιο χρειάζονται, χρειάζεται ακόμα λίγο χτένισμα έτσι ώστε να επιτευχθεί και ο στόχος που θέλετε και εσείς όπως η πλήρης ανεξαρτησία γιατί μόνον οι ειδικοί οργανισμοί που χορηγούν αυτές τις ετικέτες είναι σε θέση να κάνουν την εξέταση που πρέπει και δεν χρειάζεται ολόκληρο καινούριο σύστημα. Θα ήταν πολύ ψηλό το κόστος. Νομίζω ότι αυτά ήταν όλα κύριε Πρόεδρε, τα βασικά τουλάχιστον. Αν υπάρχει κανένα συνάδελφος που θέλει να προσθέσω τίποτα ή αν θέλετε αποσαφηνήσεις. Νομίζω όμως ότι η γενική πληροφόρηση είναι πλήρης. Ε, Σας ευχαριστώ. Ήσασταν ε, πολύ περιεκτικός για την ε, αφοσίωση της ε, Βελικής Προεδρίας σε αυτό το θέμα και την επιμέλεια με την οποία έρχεται και μας ενημερώνει. Και για την ανάμειξη στην ομάδα εργασίας. Σπάνια ακούμε κάτι τέτοιο στην Επιτροπή. Γιατί χαίρομαι που μας αφήνεται ανοιχτό αυτό το παράθυρο συνεργασίας. Και αυτό το κατάλαβαν και οι πολίτες, γιατί ε, αναμεταδίδεται απευθείας η συνεδρία της Επιτροπής και φαντάζομαι όσοι ενδιαφέρονται για την αγορά των δομικών προϊόντων θα ενθουσιαστούν με αυτό το άνοιγμα του Συμβουλίου. Ακούσαμε πολλές ε, πληροφορίες, καταρχήν το θέμα του ενιαίου σημείου επαφή ε, του point of contact και για υπηρεσίες και για προϊόντα και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα των δομικών υλικών και χρειάζονται πραγματικά τεχνικές πληροφορίες. Χαίρομαι που θα προβλεφθούν κονδύλια για αυτά τα contact points. Κυρία Στάιλερ, θέλετε μετά την παρουσίαση και του Συμβουλίου να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τον κύριο Βερτής και τον ευχαριστώ θερμά που ήρθε τελικά. Ήταν δικό μα το λάθο, γιατί έγινε αλλαγή το σημείο τη ημερήσια διάταξη και συζητήσαμε νωρίτερα το δικό μου θέμα. Πάντω, περιμένουμε με ανυπομονησία την συζήτηση που θα έχουμε αργότερα με του κοιόδη ηγητέ και με εσά. Και φυσικά, περιμένουμε την εξέταση των τροπολογιών και την ψηφοφορία τον Νοέμβριο. Σα ευχαριστώ θερμά, κυρία Στάιλερ, και ευχαριστώ και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε στη συνεδρίασή μας και μας ενημέρωσαν. Ολοκληρώνουμε το σημείο 5 και επιστρέφουμε στο σημείο 4 για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Επιτροπή με επικεφαλή τον Ανδρέας Σβάπ, τον εισηγητή μας, ε, εκπώνησε δύο εκθέσεις, ζήτησε μάλλον την εκπώνηση δύο εκθέσεων και μελετών που θα μας ε, βοηθήσουν στην κατάρτιση των εκθέσεών μας. Έχουμε μοιράσει τα αντίγραφα αυτών των δύο μελετών. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους ορισμούς, από ό,τι φαίνεται και κάποιες εκκρεμότητες στο κεφάλαιο 5, ιδιαίτερα τις γενικές συνέπειες της εναρμόνισης. Επίσης, τις διάφορες αμοιβές ευθύνες. Έχουμε τον καθηγητή Σόλτερ Νίκερ, Σόλτερ που ήταν έθερμος υποστηρικτής της Επιτροπής μας και παρόν σε πολλές δημόσιες ακροάσεις θα δώσει απάντηση στο θέμα των ορισμών στο σημείο 1 και ο κύριος ε, καθηγητής Γιάνσεν θα μας δώσει κάποια στοιχεία για το σημείο 2, την εναρμόνιση των ε, άδικων τρόπων ελέγχου. 10 λεπτά θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας. Μετά τον κύριο Σαφ, την κυρία Σαλντεμόζε, εκπροσωπεί την κυρία Κέπχαρ. Δεν ξέρω ποιος εκπροσωπήσει τους φιλελεύθερους. Η κυρία Τουρίνεν δεν έχει έρθει ακόμη. Δεν έχουμε και πολλούς σκιώδεις ε, δυστυχώς στην συνεδρίαση. Πάντως ε, θα είναι χρήσιμη η παρουσίαση από τους εμπειρογνώμονες. Θα αφιερώσουμε μία ώρα στη συζήτηση κατόπιν, αν προλάβουμε. Και επαναλαμβάνω, κύριε Σούλτε, κύριε καθηγητά Σούλτενόλ, και έχετε ένα δεκάλεπτο. Μπορείτε να ρίχνετε μια ματιά και στο χρονόμετρο. 10 λεπτά για την πρώτη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα καταρχάς. Κυρίες και κύριοι, ε, με ρωτήσατε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος πλήρως εναρμονισμένων ορισμών στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Και χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Καταρχήν, η πρώτη μου σχεδόν μονολεκτική απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα πλήρως εναρμονισμένων ορισμών. Είναι τελείως ανέφικτο και αυτό για τους εξής λόγους. Ο όρος πλήρης εναρμόνιση αφορά ένα επίπεδο προστασίας σε οδηγίες και προβλέπει τη διακριτική ευχέρεια που έχουν τα κρατη την ελευθερία που έχουν τα κρατη να καθορίσουν το δικό τους επίπεδο προστασίας. Βέβαια, οι οδηγίες σχεδόν ποτέ δεν καθορίζουν ένα επίπεδο προστασίας. Αυτό το κάνουν μόνο οι κανονισμοί. Γι' αυτό και οι οδηγίες από αυτή την άποψη του επίπεδου προστασίας είναι ουδέτερες ως προς την πληροφορία αυτή. Και μάλιστα η ερώτηση αυτή δεν είναι καθόλου χαζή, αλλά πιστεύω ότι πίσω από την ερώτηση αυτή βρίσκεται η έμεση ερώτηση αν η κοινοτική νομοθεσία μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να αντιγράψουν πιστά τους ορισμούς και τους ορισμούς της οδηγίας και τη μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία. Αν μπορούν να κάνουν μια απλή αντιγραφή και επικόλυση, δηλαδή μια πιστή αντιγραφή των ορισμών. Αυτή είναι η ουσιαστική ερώτηση. Μπορεί μια τέτοια λοιπόν οδηγία να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να κάνουν πιστή αντιγραφή των ορισμών. Όχι είναι η απάντηση. Ένα κατηγορηματικό όχι. Αν και σε ορισμένε περιπτώσει τα κράτη-μέλη έχουν εύλογου λόγου να προσαρμόσουν του δικού του ορισμού, όχι βέβαια πιστά, κατά τη μεταφορά κάποιων οδηγιών. Και μάλιστα μερικέ φορέ έχουν και συμφέρον είναι και ακόμη πιο απαιτητικά τα κράτη-μέλη. Βέβαια, μια τέτοια οδηγία πλήρω εναρμόνιση έχει αντίστοιχο αποτέλεσμα στι εθνικέ νομοθεσίε. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια γενική απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα και πάλι εξαρτάται από του συγκεκριμένου ορισμού. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Καταρχήν, γιατί ακόμη και μια, πλήρης, μια οδηγία πλήρους εναρμόνιση δεν μπορεί να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να κάνουν απλό copy-paste, μια αντιγραφή και επικόλυση των κανόνων, μια πιστή τυφλή αντιγραφή. Η απάντηση είναι απλούστατη. Το άρθρο 288 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι μια οδηγία θα είναι δεσμευτική ως προς το αποτέλεσμα που επιδιώκει και εξαρτάται από τα κράτη-μέλη, από τις εθνικές αρχές να επιλέξουν τον τύπο και τις μεθόδους για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Δηλαδή, η συνθήκη ρητά επιτρέπει στα κρατημέλη να βρουν τους τρόπους που κρίνουν σκόπιμους ε, για να υλοποιήσουν του στόχου της οδηγίας, χωρίς όμως να χρησιμοποιούν κατά ανάγκη τους ορισμούς της οδηγίας ή χρησιμοποιώντας άλλους ορισμούς. Για παράδειγμα, είναι άσχετο για το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή αν η εθνική νομοθεσία αποκαλεί τον καταναλωτή καταναλωτή ή απλώς αγοραστή ή με μία άλλη λέξη. Είναι προφανές όμως. Τα κράτη-μέλη καταρχήν είναι ελεύθερα να μην κάνουν ένα, προβούν σε ένα ορισμό της έννοιας ε, της, ε, που χρησιμοποιεί η οδηγία. Ή απλώς να χρησιμοποιήσουν τον όρο ενοχή, συμβόλαιο ή σύμβαση χωρίς να τον προσδιορίζουν. Ή να χρησιμοποιήσουν άλλες τεχνικές ορισμού που δεν είναι οι συνηθισμένες με βάση τον αριστοτελικό τύπο. Δεν θα σας εξηγήσω τώρα πώς λειτουργεί η λογική, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλες τεχνικές. Τα κράτη-μέλη καταρχήν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλες λέξεις ή φράσεις που χρήζουν ε, ορισμού. Για παράδειγμα, μπορούν να πούν αντί για καταναλωτής ο τελικός παραλήπτης ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία, έναν ορισμό, να διαλέξουν έναν ορισμό από την οδηγία, αλλά να του προσθέσουν άλλο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορούν να, χρησιμοποιήσουν, να περιλάβουν και τα νομικά πρόσωπα στην έννοια του καταναλωτή, στην εθνική του νομοθεσία, κάποια κρατημέλη, αν το επιθυμούν. Παρ' όλα αυτά, η οδηγία πλήρου εναρμόνιση και οι ορισμοί μια τέτοια οδηγία πλήρου εναρμόνιση θα έχει αντίκτυπο στι εθνικέ νομοθεσίε. Και ο αντίκτυπος αυτός εξαρτάται από, τις, από τους συγκεκριμένους ορισμούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες ορισμών σε αυτό το σχέδιο οδηγίας, αλλά και γενικώ σε όλα τα σχέδια οδηγιών. Για παράδειγμα, η πρώτη κατηγορία είναι ορισμοί που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογή. Που χρησιμοποιούνται δηλαδή σε κανόνε που προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογή του ορισμού. Και το απλούστερο παράδειγμα είναι ο όρο καταναλωτή γιατί η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτή ισχύει μόνο για τους καταναλωτές. Τέτοιου είδους ορισμοί επιτρέπουν στα κράτη-μέλη τουλάχιστον να διευρύνουν αυτόν τον ορισμό, να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής, την εμβέλεια του ορισμού. Γιατί ακόμη και πέρα μιας οδηγίας πλήρους αναρμόνησης μπορούν τα κρατη να διευρύνουν την εμβέλεια ενός ορισμού. γιατί συνήθως η πλήρης εναρμόνιση αφορά το πεδίο εφαρμογή οδηγία. Αλλά πέραν του πεδίου εφαρμογή, το κράτος μέλο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά δεσμεύεται από τη συνθήκη και άλλε υποχρεωτικές και νοητικέ διατάξει. Τα κράτη-μέλη δηλαδή μπορούν να προστατεύσουν και μη καταναλωτές. Νομικά πρόσωπα, για παράδειγμα. ένα μικρό συνεταιρισμό, για παράδειγμα. Μια μικρή ένωση, ένα μικρό σωματείο. Να του χαρακτηρίσουν είτε να του χαρακτηρίσουν καταναλωτέ, είτε ακόμη και να του χαρακτηρίσουν καταναλωτές, να επεκτείνουν την προστασία και σε αυτού. Η άλλη κατηγορία είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Αν έχουμε μια οδηγία πλήρου εναρμόνιση, τα κράτη-μέλη καταρχήν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στενότερο ορισμό, συσταλτικότερο ορισμό του καταναλωτή. Αυτό καταρχήν ισχύει, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσει. Αν ένα κράτο καταφέρει να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας με πιο στενό ορισμό μπορεί να το κάνει. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ε, τον κανόνα οι γάτε θεωρούνται σκύλοι, ας πούμε. Και ως προς τις συμβάσεις, πολλές χώρες χρησιμοποιούν διαφορετική έννοια για την σύμβαση υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μια σύμβαση έργου μπορεί να θεωρηθεί για τους σκοπούς της οδηγίας ως σύμβαση υπηρεσίας, παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει νομικός λόγος που να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν πιστά τον, τον, ορισμό. Άλλη κατηγορία ε, ορισμών είναι οι ορισμοί που αφορούν ένα επίπεδο προστασίας, mm. που δεν καθορίζουν το, την εμβέλεια, το πεδίο εφαρμογή του ορισμού, αλλά το επίπεδο προστασία του ορισμού. Εδώ τα κράτη-μέλη έχουν λιγότερη διακριτική ευχέρεια. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται σε ένα durable medium, σε ένα μέσο που θα έχει μια αντοχή, μια διάρκεια. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν διαφορετικό ορισμό, όχι το durable medium, αλλά θα είναι δύσκολο να του δώσουν διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί το durable medium λέει τι θα πρέπει να γίνεται για να ενημερωθεί ο καταναλωτής. Η τρίτη κατηγορία ορισμών είναι οι ορισμοί που αφορούν την, τον τύπο, τον στάνταρ τύπο της οδηγίας. Και εδώ, στόχος της οδηγίας είναι τέτοιοι ορισμοί, standard form relevant, που χρησιμοποιούνται και στους, ε, στα έντυπα που δίνονται στο παράρτημα της ε, οδηγίας, μπορούν και μάλιστα ο κοινοτικός νομοθέτης μπορεί ακόμη και μέσω μιας οδηγίας να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το έντυπο που προβλέπει η οδηγία. Το στάνταρ έντυπο. Mm. Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να αντιγράψουν πιστά αυτά, το, αυτά τα έγγραφα, αυτά τα έντυπα. Ως προς, την, ως προς τον τύπο δηλαδή, ως προς το έντυπο, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα. Και αν είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο έντυπο, ένα τέτοιο τύπο, ίσως χρειαστούν και άλλες προσαρμογές των ορισμών τους για να αποφευθούν αντιφάσεις στην εσωτερική τους νομοθεσία μπορεί να, να εξαναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν τον καταναλωτή, καταναλωτή στο έντυπο για παράδειγμα. Οπότε αν στο έντυπο αναφέρεται ο όρος καταναλωτής, δεν μπορούν σε άλλα τμήματα της εσωτερικής νομοθεσίας να χρησιμοποιούν διαφορετικό ορισμό ή διαφορετική... διαφορετικό όρο. Προχωρώ στην σύνοψή μου. Οδηγίες πλήρους εναρμόνισης που χρησιμοποιούν ορισμούς θα έχουν περιορισμένες επιπτώσεις, περιορισμένο αντίκτυπο στην εσωτερική νομοθεσία ενός κράτους μέλους και άρα και στην εσωτερική αγορά. Και το πιο ενοποιητικό αποτέλεσμα οι ορισμοί θα το έχουν σε αυτά τα έντυπα, στις, στα, στάνταρ, στα στάνταρ έντυπα. Επίσης, ίσως ήταν χρήσιμο η κοινοτική νομοθεσία να προβλέπει ότι ο νομοθέτης χρησιμοποιεί, δημιουργεί κάτι ενοποιημένα καλό για τους καταναλωτές. Και αυτό θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε EU Model Withdrawal Form, τονίζοντας ότι είναι κάτι καλό για τον καταναλωτή. Στην Ανταλουσία, για παράδειγμα, έχουμε αυτές τις γαλάζιες σημαίες Αυτά, ευχαριστώ. Well, thank you very uh, Ευχαριστούμε πολύ για τη σαφέστατη αυτή παρουσίαση τόσο απλή. Το τελευταίο που είπατε είναι κάτι το οποίο ήδη το λάβαμε υπόψη μας στην οδηγία Time Share όπου είχαμε προτείνει μεταξύ άλλων προτύπων και ένα σαν το δικό σας και το δέχτηκε και το Συμβούλιο. Είναι λοιπόν θέματα που πρέπει να τα δούμε και στα πλαίσια αυτής της πρότασης για τα δικαιώματα των καταναλωτών και καταναλωτριών. Λοιπόν, οι ερωτήσεις αργότερα. Τώρα ο καθηγητής Γιάνσεν που θα μας μιλήσει για τους όρους των διαφόρων συμβολέων και πάλι για την εναρμόνιση που θα είναι το κοινό στοιχείο σε όλες τις παρουσιάσεις. Και εσείς δέκα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά την παρουσίαση της μελέτης μας θα είμαι πολύ σύντομος να σας παρουσιάσω τέσσερα μοντέλα για την εναρμόνιση του ελέγχου. Και για κάθε μοντέλο έχω και μία διαφάνεια. Ναι, συγγνώμη, θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε, να μου δείξετε όλες τις διαφάνειες. Αυτή η πλήρης εναρμόνιση δεν θα σήμαινε ότι οι φορείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν σε όρους σε όλη την Ευρώπη. Στις αρχές του έτους ε, δημοσίευσα ένα άρθρο για το πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό και πώς θα έπρεπε να ε, αλλάξει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προκειμένου οι φορείς να μπορούν να εφαρμόζουν τους ίδιους όρους σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα, μάλλον ο λόγος που θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, είναι ότι είναι καλό όχι μόνο για τους εμπορευομένους, αλλά προκειμένου να υπάρχει ενιαία συμβατική νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα υπάρχει, για παράδειγμα, μάλλον δεν γίνεται να υπάρχει ενιαίος έλεγχο χωρίς να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ενιαία συμβατική νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών, θα προσπαθήσω να το πετύχω αυτό μέσα μέσω των καταχρηστικών ε, ρήτρων. αλλά αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο συμβατικό δίκαιο όλων των κρατών μελών. Και γι' αυτό λοιπόν θα προαπαιτούσε τεράστιες αλλαγές στο τρέχον κεφάλαιο 5. Γιατί οι σχετικοί κανόνες είναι μικρό τμήμα των κανόνων που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τον έλεγχο των αθέμπτων συμβάσεων. Και μάλιστα αυτοί οι κανόνες υφίσταντο και πριν την οδηγία την Ευρωπαϊκή του 1993 και πρώτου δημιουργηθούν τα συγκεκριμένα μέσα ελέγχου. Τα συγκεκριμένα μέσα αυτά πλέον αποτελούν ένα μόνο τμήμα του ελέγχου. Αυτό τι σημαίνει ότι θα έπρεπε να αντικατασταθεί μεγάλο τμήμα των ενοχικών, του ενοχικού δικαίου των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους όρους αυτούς. Και αυτό με τη σειρά του ασφαλώς συνεπάγεται ότι θα έπρεπε να ανατεθεί στο, Ευρωπαϊκό, ε, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η ανάπτυξη του ενοχικού δικαίου. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα καταλήγουν στο δικαστήριο. Πιο πολλές συμβάσεις σήμερα αποτελούν ε, τυποποιημένες συμβάσεις. Άρα το ΔΕΚ θα έπρεπε τελικά να έχει τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις αυτές. Θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε και θεσμικού τύπου αλλαγές δεν νομίζω ότι αυτό τίθεται, τίθεται τέτοιο θέμα σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν ως ακαδημαϊκή κοινότητα δεν μπορούμε να το συστήσουμε αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για αυτά που είπα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο θεμητών ή μη θεμητών συμβάσεων. Έχουμε για παράδειγμα κανόνες ε, σε ό,τι αφορά τις ε, καταναλωτικές πιστώσεις. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες ε, ακύρωσης των πιστώσεων αυτών. Αυτό δεν είναι σαφές αν θα μπορούσε να συνεχίσει να υφίσταται υπό το αναθεωρημένο κεφάλαιο 5, εναρμονισμένο δηλαδή. γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι τέτοιοι κανόνε στη Γερμανία και νομίζω ότι σε όλα τα νομικά συστήματα υπάρχει κάποιο σύστημα ελέγχου των τιμών. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν ε, παρόμοιοι κανόνε που να προβλέπουν, αν δεν προβλέπονται παρόμοιες διατάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρη εναρμόνιση. Μια επίσημη πλήρη εναρμόνιση. Θα είμαι σύντομο γιατί πολλά ακούσατε και τον προηγούμενο ομιλητή. Η ιδέα ποια είναι να εφαρμοστεί μια παρόμοια ορολογία στα κράτη-μέλη. Να πούμε λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους όρους. Αν όμως είναι διαφορετική η ερμηνεία των όρων, αυτό τι θα σημαίνει στην πράξη, ότι δεν θα υπήρχε καμία διαφορά με τη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση. Αλλά δεν θα λειτουργούσε το μοντέλο αυτό, γιατί θα υπήρχαν παρανοήσεις και νομικές ε, διαφωνίες. Καταστροφή θα σήμαινε αυτό σε νομικό επίπεδο. Αν, αν χρησιμοποιήσαμε τους ίδιους όρους για διαφορετικά πράγματα. Οι νομικοί θα είχαν δυσκολία να κατανοήσουν τα διαφορετικά ε, νομικά συστήματα και κανείς δεν θα καταλάβαινε τελικά τι σημαίνει αυτή η πλήρης εναρμόνωση. Τα ίδια αποτελέσματα, την ίδια ορολογία. Όχι. Και νομίζω ότι αναγκαστικά θα καταλήγαμε σε μια μη ίση αντιμετώπιση των πολιτών. Αυτό θα ήταν η συνέπεια. Και αυτό τι σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλήρως εναρμονισμένους καταλόγους μαύρους, μαύρες λίστες, γκρίζες λίστες ε, τέτοιων, ε, για τέτοιες ρήτρε. Γιατί τα δικαστήρια που εφαρμόζουν τις ε, γενικές ρήτρε, πολύ απλά πάντα έχουν τέτοιες γκρίζες ή μαύρες λίστες δικές τους. Στην επόμενη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση. Πλήρη εναρμόνιση η οποία θα περιοριζόταν σε κάποιες πτυχές του κεφαλαίου 5. Πέρα από τη δοκιμή αυτή θεμητότητας. Συζητήσαμε θέματα εφαρμογής της δοκιμής αυτής θεωρητικά θα ήταν δυνατόν, αλλά τα αποτελέσματα στην πράξη δεν θα ήταν καλά. Δεν θα βοηθούσαν τους ε, εμπορευομένους και τους υπόλοιπους φορείς ή τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της ενιαίας της ιστορικής αγοράς. Δεν θα χρησιμοποιούνταν ενιαίοι όροι τυποποίησης, δεν θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αυτό οι καταναλωτές. Και θεωρώ ότι μια τέτοια εναρμόνιση θα προκαλούσε μάλλον μια αθέμητη αθέμητα περίπλοκη κατάσταση. Άρα μπορεί από τεχνική άποψη να φαίνεται εφικτό αυτό, δεν μπορούμε όμως να το συστήσουμε παρόλα αυτά. Γιατί ε, προκαλεί άχθος χωρίς να έχει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Ένα πιο γενικό σχόλιο τώρα για την στοχοθετημένη αυτή προσέγγιση. Νομίζουμε ότι πολύ πιο καλό θα ήταν να εφαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο θεσμό, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα απόσυρσης. Εκεί θα είχε νόημα, αλλά όχι σε ένα γενικό κανόνα. Γιατί εκεί δεν θα είχε πιο θετικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, θα προκαλούσε νομικές δυσκολίες και κάθε νομικό πρόβλημα έχει επιπτώσεις και στον καταναλωτή. Γιατί θα προκαλέσει νομική επιβεβαιότητα. Άρα τη συστήνουμε τελικά, μία ελάχιστη εναρμόνιση στην επόμενη διαφάνεια. Δηλαδή, στοχτατημένη εναρμόνιση από άλλα κεφάλαια. Οι επιπτώσεις θα ήταν οι εξής οι καταναλωτές ε, θα μπορούσαν να υπολογίζουν και να βασίζονται σε λίγο πολύ ίδιους όρους ε, ενοχικούς. Και πολύ απλά πιστεύω ότι στην παρούσα φάση οτιδήποτε άλλο είναι εντελώς ανέφικτο. Και ακόμα και αν υπήρχαν τυποποιημένοι όροι, θα χρειαζόταν μετάφραση και η μετάφραση θα προαπαιτούσε νομικό έλεγχο. Άρα και να είχαμε εναρμόνιση πάλι δεν θα μπορούσαμε να εξαφταθούμε τους νομικούς. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας παρουσιάσω σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Τώρα σε ό,τι αφορά το επίπεδο εφαρμογή μάλλον για την προστασία των επιχειρήσεων και των ε, άλλων φορέων, των μη καταναλωτών. Δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε τα κράτη-μέλη από το να επεκτείνουν την προστασία αυτή και σε άλλους μη καταναλωτέ. Γιατί πολύ απλά δεν έχει νομική αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μεγάλη παρανόηση αναφορικά με το άρθρο 3, παράγραφο 1 τη πρότασης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε ότι ίσως να χρειαστεί κάποια διευκρίνηση, κάποια ε, επεξήγηση στο άρθρο 4 των τελογικών σκέψεων. Σας ευχαριστώ. Thank you Και εμείς σας ευχαριστούμε <laughs> για την σαφέστατη και αυτή παρουσίαση. Υπάρχουν και αντίγραφα εδώ για όποιον ενδιαφέρεται της παρουσίασης. Πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά για την καθοδήγηση των εργασιών μας υπό την ησυγεσία του κυρίου Σβάμπ. Δεν ζητούμε μέγιστη εναρμόνιση, αλλά θέλουμε να ταυτίσουμε τα θέματα στα οποία θα έπρεπε να υπάρξει εναρμόνιση. Καλό τώρα λοιπόν τον εισηγητή κύριο Σβάμπ να αρχίσει τη συζήτηση. Και φαντάζομαι και άλλοι θα θέλουν να μιλήσουν. Όποιος θέλει να το ζητήσει. Και αν θέλουν και οι ομιλητές να σχολιάσουν. Ο κύριος Βάμπα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο καθηγητές που μας παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε ό,τι αφορά τις παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον καθηγητή Γιάνσεν και από τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του για το άρθρο 5 και το τι θα συνεπαγόταν ε, εναρμόνιση σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, το κεφάλαιο 5. Πιστεύω ότι γενικά οι αμφιβολίες που εκφράσατε είναι πολύ εύλογες σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα προέκυπταν όλα αυτά τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τον αναστικό κώδικα. Γι' αυτό να ομολογήσω ανοιχτά ότι γνωρίζω ότι από επιστημονική αποψή είστε πολύ πιο καταρτισμένος, ωστόσο στην πράξη θεωρώ ότι θα ήταν πιο αισιόδοξη η κατάσταση. Δικαίως είπατε ότι η εναρμόνιση των κανόνων τελικά θα ήταν ο πιο σωστός τρόπος για το Ευρωπαϊκό Ενοχικό Δίκαιο και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των 27 νομικών συστημάτων των κρατών μελών δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα επιπλέον ε, σύστημα, γιατί θεωρώ ότι η Ευρώπη της ενοποίησης έχει να παρουσιάσει πολύ, πολύ πιο πολλά πλεονεκτήματα από μια διακυβερνητική Ευρώπη. Αλλά σωστά είπατε ότι ο δόμος αυτός θα είναι πολύ οδυνηρός και πολύ μακρύς για και χαίρομαι που είπατε ότι το κεφάλαιο 2 και 3 ως πλήρως εναρμονισμένα κεφάλαια θα λειτουργήσουν άψογα, γιατί αυτό αποτελούσε ένα ερώτημα, ένα θέμα της Επιτροπής και συμφωνώ όταν λέτε ότι το, στο κεφάλαιο 4 η πλήρης εναρμόνιση θα είναι πιο δύσκολη, αλλά όχι μόνο λόγω της διαφάνειας για τις επιχειρήσεις, αλλά για να διευκολύνουμε την νομική προσέγγιση επιλέξαμε τον δρόμο αυτό και μας παρουσιάσατε σαφέστατα ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα και ποια θα ήταν τα μειονεκτήματα μια ελάχιστη ή μια πλήρου εναρμόνιση. Αναφέρατε not recommended, ε, δεν συστήνεται, αλλά αν σας ρωτούσα ποιον από τους δύο δρόμους θα ακολουθούσατε αν σας αναγκασμένο να, να, να επιλέξετε ένα από τους δύο, θα με ενδιαφέρει να ακούσω ποια είναι η απάντηση. Και τέλος, ε, Χαίρομαι που αναφέρθηκατε στο θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Και εσείς το είπατε αυτό, κύριε Όλκεν, και νομίζω ότι καταφέραμε ό,τι θέλαμε να πετύχουμε για το κεφάλαιο 1. Δεν μιλώ για πλήρη εναρμόνιση, μιλώ για την ενιαία διαμόρφωση η οποία δεν θα πρέπει πλέον να αποτρέπει την προστασία και φορέων πέρα των καταναλωτών. Γιατί αυτό συχνά μας ανησυχεί. Απασχολεί πάρα πολύ τα κράτη-μέλη, ότι θα, ότι θα περιορίζονται ε, αν θέλετε, σε περίπτωση που θα εναρμονιστούν οι όροι στο κεφάλαιο ένα σε ό,τι αφορά την προστασία πέρα των καταναλωτών. Γιατί υπάρχει και η σκέψη αυτή. Εφόσον είναι τόσο θετικά τα αποτελέσματα, γιατί χρησιμοποιώντας αυτούς τους απλοποιημένους ορισμούς σε άλλους τομείς, ε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε μεγαλύτερη νομική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν ε, συμφωνώ ότι θα ήταν πολύ καλή αυτή η απλοποίηση. Θεωρείτε ότι η απλοποίηση αυτή θα ήταν ωφέλιμη χωρίς να συνεπάγεται αν θέλετε, άχθος και βάρος για τα κράτη-μέλη. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που ήθελα να θέσω. Ευχαριστώ, κύριε Σαλτεμόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώ ε, δεν με καταλαβαίνουν πολύ όταν μιλώ τη γλώσσα μου, αλλά θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, παρακαλώ να σα ε, σας ευχαριστώ μάλλον για τι δύο εξαιρετικέ αυτέ παρουσιάσει. ιδιαίτερα για τα συμπεράσματά σα. Είστε Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και στη διαδικασία που ξέρουμε, που έχουμε γνωρίσει, μπορέσατε να μας εξηγήσετε καθαρά ποια θα ήταν τα ωφέλη από μία εναρμόνιση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την υποστήριξή σας. Αλλά πρέπει και να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τις συστάσεις του κυρίου Σβάμπ. Βέβαια θα επανέλθω και στους ορισμούς, ε, απλώς για να είμαι βέβαιη ότι κατάλαβα καλά. Καλά, μας είπατε ότι ακόμη και αν υπάρξει πλήρης εναρμόνιση των ορισμών, ούτως ή άλλως δεν θα είναι ενιαία η ερμηνεία τους σε όλα τα κράτη-μέλη. Καλά το κατάλαβα. Δηλαδή τότε, σε αυτή την περίπτωση, γιατί να κάνουμε καν εναρμονισμένους ορισμούς αφού η ερμηνεία τους θα είναι ούτως ή άλλως διαφορετική ανακράτος μέλος. Γιατί. Για ποιο λόγο διαπίανε τι Παρακαλώ. Γιατί να κάνουμε αυτόν τον κόπο αφού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να, να τα ξυλώσει αυτά που θα έχουμε πλέξει εμείς. Γιατί χρειάζεται ευρωπαϊκό έγγραφο, ευρωπαϊκό πρότυπο αφού δεν θα είναι πανευρωπαϊκή εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε και αυτό είναι το μόνο ερώτημα που είχα να θέσω. Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως κανένα συνάδελφος θέλει να θέσει κανένα άλλο ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Σμιτ. Δεν είμαι σκιώδης. Ήμουν σκιώδης στην Επιτροπή Εικόν, αλλά πρέπει να πω ότι πάντοτε ήμουν υπέρ της πλήρους εναρμόνισης για την πληροφόρηση των καταναλωτών και καταναλωτριών. Διότι μόνο δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να υπάρχει λειτουργούσα ενιαία αγορά. Ερωτώ λοιπόν τα εξή. Τι θα χάσουμε αν εφαρμόσουμε αυτά που ζητάτε. Πρέπει να υπάρχει κάποιο τίμημα μάλλον. για να μην λειτουργήσει πλήρως η εσωτερική αγορά. Ποιο είναι το τίμημα. Να μας πείτε λίγο παραπάνω γιατί εσείς μας συστήσατε να μην κινηθούμε πολύ γρήγορα λέει γιατί είναι τεράστια τα προβλήματα κτλ. Ενώ τα τελευταία 10-15 χρόνια αυτό ακριβώς πράταμε. Θα ακούσω με μεγάλη προσοχή τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κανείς άλλος. Εγώ να θέσω ένα. Νομίζω προς τον κύριο Γιάννησεν, αλλά ίσως να αφορά και τους δύο. Όταν αναφέρατε μερικά από τα προβλήματα των ενιαίων προτύπων, είχατε πει ότι θα μπορούσαν να λυθούν από ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, το οποίο επεξεργαζόμαστε όμως όπως θα ξέρετε. Και βέβαια και από τη νομική επιτροπή ξέρουμε και τις τροπολογίες της ότι κάτι τέτοιο αναμένουν το ενιαίο πλαίσιο δηλαδή. Τι φρονείτε, γιατί εδώ υπονοείται ότι αναγνωρίζετε ότι καλό θα ήταν να υπάρξει ένα τέτοιο ενίο πλαίσιο αναφοράς το οποίο ακριβώς όπως είπα και πριν άλλες δύο φορές επεξεργαζόμαστε. Αν και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, υπάρχει κάποια έλλειψη ενιαία στρατηγικής προσέγγισης, αλλά αυτό. Α, και η κυρία Στάιλερ ήθελε. Αν δεν απατώμε θα σας δώσουμε το λόγο. Αλλά και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι εδώ. Πρώτα η κυρία Στάιλερ και μετά εσείς. Ευχαριστώ πρόεδρε και τους εισηγητάς, τους προγνώμονες. Συμφωνώ με την κυρία Σάλντεμος για το θέμα της πλήρους εναρμόνισης, αλλά την περασμένη εβδομάδα φάνηκε, γιατί και εσείς είστε νομομαθείς, ότι τίθεται το ερώτημα, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επαρκής τρόπος εφαρμογής των υπαρχόντων κανόνων για τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες γιατί προβλέπονται και περικοπές στους προϋπολογισμούς τουλάχιστον των κρατών μελών και μια οργάνωση καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό. Αν οι καταναλωτές έχουν σαφή και ρητά δικαιώματα Ξέρουμε ότι δεν είναι τέλειος ο κόσμος βέβαια, αλλά στις εκλογικές μας περιφέρειες μειώνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μήπως πρέπει να συμβιβαστούμε λοιπόν μεταξύ αυτών που θέλουμε και αυτών που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Αν είχατε ένα λευκό χαρτί μπροστά σας, τι θα προτείνατε. Α, εδώ μπορεί να χρειαστεί ολόκληρη νύχτα για να απαντήσουν. Λοιπόν, τώρα που με βλέπετε στο ηλιόφως δεν μπορώ να σας δω εγώ. Λοιπόν, κύριε Πέτρη θέλετε να κάνετε κανένα σχόλιο και μετά οι καθηγητέ. Ευχαριστώ. Um, Καταρχήν για τους στερεότυπους όρους των συμβάσεων γιατί το θέμα των ορισμών εμένουμε σε αυτά που λέμε στους ε, ορισμούς, για τους ορισμούς στην πρόταση. Σε ό,τι αφορά τους αθέμητους όρους, η πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να σας δείξουμε την πρόθεσή μας ε, που κρύβεται πίσω από αυτήν την εναρμόνιση. πρόθεσή μας λοιπόν είναι να έχουμε μια ασθενέστερη με εναρμόνιση, αλλά πιο στοχοθετημένη. Δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε τους ε, υποχρεωτικούς όρους του ενοχικού δικαίου, τους εθνικούς που ισχύουν για συγκεκριμένες ε, συμβάσεις, όπως είναι τα, οι ασφαλιστικές συμβάσεις. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Απλώς ε, θέλησαμε μια ελάχιστη εναρμόνιση για τους ενοχικούς όρους των συμβάσεων. Επίσης, δεν ήταν πρόθεσή μας να κρίνουμε με, τους ίδιους, με τον ίδιο τρόπο τους όρους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καταρχήν είναι ανέφικτο. Θα ήταν ανέφικτο ακόμη και να έχουμε πλήρη εναρμόνιση τη, του τεστ α, αθεμητότητας. Γιατί τα κράτη-μέλη ερμηνεύουν διαφορετικά πολλές φορέ του όρου, του ενοχικούς ανάλογα με την εθνική νομοθεσία ή τις ε, εμπορικέ πρακτικές. Για παράδειγμα, το δίκαιο ε, σε ό,τι αφορά την εκμίσθωση, το βάρος αποζημίωσης ε, για, για τις ζημιές που γίνονται στο μίσθωμα, επιβαρύνει στο Βέλγιο τον ε, μισθωτή, ενώ στη Γερμανία, για παράδειγμα, τον εκμισθωτή, τον ιδιοκτήτη. Επίσης, ε, αν δεν είναι αυτή η πρόθεση, τι επιδιώκει πλήρη εναρμόνιση. Το σημαντικό είναι εδώ να αντιληφθούμε ότι αυτό που επιδιώκουμε είναι να βελτιώσουμε μία κατάσταση εξάντε αξιολόγησης των ε, ενοχικών όρων. Δεν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σε περίπτωση έναρξης της αντιδικίας, όταν δηλαδή υπάρχει μια αμφισβήτηση των ε, συμβατικών όρων. Ή αν υπάρξουν διαφορές ερμηνείας μεταξύ των δικαστηρίων σε περίπτωση αντιδικίας. Ούτε αυτή την κατάσταση πρόκειται να τη βελτιώσουμε με χάρη στην εναρμόνιση. Άλλωστε και οι επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά θα ήταν ελάχιστες. Γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός των καταναλλακτικών συμβάσεων που καταλήγουν σε αντιδικία. Και ακόμη μικρότερος είναι ο αριθμός των συμβάσεων που καταλήγουν στο δικαστήριο. Στα εθνικά δικαστήρια. Οπότε είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι μέσω της εναρμόνισης προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τον ε, συμβαλόμενο για τον έμπορο να προσδιορίσει εκ των προτέρων κάποιους συμβατικούς ενοχικούς όρους. Τώρα, ως προς την κατάσταση στο Συμβούλιο, στις εξελίξεις στο Συμβούλιο, θα ήθελα να πω ότι εκεί επειδή έχουμε πλήρη εναρμόνιση τουλάχιστον αυτού του unfairness test, του τεστ για την διευκρινήση, για την ε, προσδιορισμό το κατά πόσο είναι αθέμητη μια σύμβαση. Αυτό το τεστ πάντως για την εξακρίβωση της, του θεμητού χαρακτήρα, του χαρακτήρα, εκεί τα κράτη-μέλη επιδιώκουν πλήρη εναρμόνιση. Και αυτό ισχύει και για τα εθνικά δικαστήρια που θα εφαρμόσουν τους κανόνες, αλλά και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης φαίνεται ότι είναι υπέρ αυτής της ε, πλήρους εναρμόνισης αυτού του τεστ εξακρίβωσης ε, του αθέμητου χαρακτήρα. Οπότε θα ήθελα και η δική σε επιτροπή να εμείνει σε αυτή την προσπάθεια επίτευξη πρόοδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εκεί συνήθω ε, τα κράτη-μέλη είναι πιο απρόθυμα ως προς την εναρμόνιση. Αλλά ακόμη και τα κράτη-μέλη εδώ είναι υπέρ τη εναρμόνιση τουλάχιστον αυτού του τεστ για την εξακρίβωση του αθέμητου χαρακτήρα. Θα δώσω τώρα το λόγο στου ε, εμπειρογνώμονε μα για μια σύντομη απάντηση γιατί σε 5-6 λεπτά πρέπει να τελειώσουμε για να περάσουμε στην επόμενη έκθεση που είναι για τους κυρίες Βάιλερ. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Κύριε Σβάπ. Για τον ενιαίο χαρακτήρα των ε, όρων. Ναι, μεν. Πιστεύω ότι είναι ως τοχοθέτηση άψογη, γιατί αυτό θα οδηγούσε στο σχηματισμό ενιαίων νήσων, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό που λέω το εξή. Με την οδηγία δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί. Γιατί αυτό που θα μας ε, βοηθούσε να καταλήξουμε στην μεγαλύτερη ενοποίηση θα ήταν αυτά τα έντυπα, τα υποδειγματικά έντυπα, τα υποδείγματα για τους κοινού όρους. το θέμα του ε, ελέγχου αθέμη του χαρακτήρα στο κεφάλαιο 4 ή 5 στην οδηγία. Να πω δύο λόγια γι' αυτό. Ήδη σήμερα τα πιο πολλά κράτη-μέλη κάνουν copy-paste, αντιγραφή και επικόλληση και κάνουν παρόμοιο έλεγχο και έχουν εντάξει στην ε, νομοθεσία τους παρόμοιους ελέγχους. Αυτό θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω αν διαφωνεί ο κ. Γιάνσεν. Και αυτό αποτελεί μία πρόοδο. Αν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να αναγκάσουμε όλα τα κρατημέλη να το κάνουν αυτό. Γιατί αν τεθεί ο στόχο η πλήρη συναρμόνιση ίσω να προσεγγίσουμε πιο πολύ τον στέχο αυτό. Γιατί σήμερα τι γίνεται. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εξέδωσε μια σχετική απόφαση που θα την γνωρίζετε που δεν μπορεί να κρίνει τις ρήτρες μη θέμη του χαρακτήρα αυτού. Μόνο αν αλλάξει η νομολογία αυτή θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια βαθιά αλλαγή στην ε, νομοθεσία των κρατών μελών. Τώρα, για μια σκέψη που φαίνεται να επικρατεί ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους, τους ίδιους ε, εμπορικού όρους σε όλη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, γιατί οι γενικοί εμπορικοί όροι πάντα ε, καταρτίζονται κατά μιας κατάστασης. Γιατί δημιουργούνται νέοι κανόνες, γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι ε, με την προηγούμενη κατάσταση. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο εκμιστοτής είναι αυτός ο οποίος ε, καταβάλει το κόστος ε, αποζημίωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να αναποιήσουμε αυτούς τους κανόνες και πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτό σε μια χώρα η οποία για παράδειγμα ε, ορίζεται ότι ο μισθωτή είναι αυτό ο οποίο είναι υπεύθυνο. Αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι αυτή οι γενικοί όροι, πέρα από κάποιε περιορισμένε εξαιρέσει, ε, έχουν γραφτεί για μια συγκεκριμένη νομική πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν με τα μέσα τα οποία συζητάμε εδώ και τώρα σήμερα, μια οδηγία δηλαδή, η οποία άπτεται και μέλλον που δεν είναι εναρμονισμένοι Και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε, κύριε Γιάνσεν, ότι δεν έχει διαφορά αν μιλήσουμε για πλήρη εναρμόνιση ή για ελάχιστη εναρμόνιση, γιατί η πλήρης εναρμόνιση ίσως να έχει το ελάχιστο πλεονέκτημα ότι θα εξανάγκαζε κάπως τα κρατημένη και θα ήταν πιο συγκρίσιμα τα πράγματα. Αλλά για να είμαι σαφής και νομίζω ότι η κυρία Στάιλερ ε, το έθιξε το θέμα αυτό, ε, έστω ότι είχαμε μπροστά μας μία κοινή σελίδα. Η οδηγία αυτή σε ό,τι αφορά την πλήρη εναρμόνιση των υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις των υποχρεώσεων παροχή πληροφοριών από επιχειρήσει και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ανάκληση είναι μια χαρά. Αποτελεί μια τεράστια πρόοδο σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Κατά τα άλλα, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και από πολιτική άποψη θέματα ε, πλήρου εναρμόνιση. Τίθεται και το θέμα των ορισμών που ανέφερα γιατί με την οδηγία αυτή δεν πρόκειται να πετύχουμε να πετύχουμε για παράδειγμα ενιαίους εμπορικού όρους για το ηλεκτρονικό εμπόριο για παράδειγμα στην Ευρώπη και άρα το ερώτημα, το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να καταρτήσουμε άλλες οδηγίες πλήρους εναρμόνισης και κατά πόσον θα υπάρξει και πολιτική αντίδραση. Και ποια είναι η εναλλακτική λύση αυτά που συμβαίνουν σήμερα με την ομάδα εργασία, να προσπαθήσουμε δηλαδή με το 28ο Καθεστώ, όπω αναφέρεται, πιο στοχοθετημένα, με ελάχιστη παρέμβαση αν θέλετε, να επιλύσουμε το θέμα. Δεν ξέρω φυσικά αν θα στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημα αυτό. Υπάρχει αυτό το μοντέλο επιπέδων. Δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρξει κοινωτική νομοθεσία. Αλλά η οδηγία αυτή θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα. Δεν πρόκειται να καλύψει όλα όσα είναι απαραίτητα. Διακόπτω στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάνσαν, χωρίς να έχω απαντήσει ωστόσο άλλα τα ερωτήματα. No, thank you very much indeed. Uh, no, we... Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε δυστυχώς και πολύ χρόνο. Πάντως ευχαριστώ για την ενθουσιώδη σας απάντηση. Κύριε Γιάννησεν, θα μπορούσατε να σχολιάσετε άλλα σημεία και κατά προτίμηση να είστε και λακωνικός. Λοιπόν. Σε λίγο θα πρέπει να αλλάξω θέση, γιατί ούτε και εσείς θα με βλέπετε όταν θα σας κάνω μήνυμα, νόημα. Να απαντήσω στον κύριο Σβάπ στα γερμανικά. Ναι, δεν μπορούμε ναι, να τα συγκρίνουμε αυτά σε ό,τι αφορά το αστικό δίκαιο, τον αστικό κώδικα. Γιατί δεν συμβαίνουν στο 10 όσα συνέβαιναν τότε. Και προφανώς εξαρτάται από την ομολογία. Απορρίφθηκε τέτοια εναρμόνιση των γενικών ρήτρων και η παρέμβαση στο εθνικό δίκαιο επειδή δεν υπήρξαν οι απαραίτητοι πόροι. Δεν ήταν θέμα αρμοδιότητα. Πολύ απλά δεν είναι εφικτό έτσι όπως έχει το ΔΕΚ σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστό σύστημα και εδώ πέρα διαφωνώ με τον συναδελφό μου. Γιατί δεν συστήνω αυτές τις λύσεις, γιατί αν σας έλεγα, μάλλον, αν είχαμε παραπάνω από δύο μήνε μπορεί να σας σύστηνα να ξαναγράψουμε το κεφάλαιο 5, γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε πάρα πολλά σημεία. Και για να απαντήσω στον Πρόεδρο, αυτό τι σημαίνει ότι ο έλεγχο των μη θεμητών όρων θα έπρεπε να τεθεί και οι τυποποιημένοι όροι θα έπρεπε να τεθούν στο ΔΕΚ. Αυτό είναι ούσια το έγγραφο. τα δικαστήρια θα χρειάζονταν κάποια τεκμηρίωση, κάποια έγγραφα αναφορά. Το θέμα είναι ότι οι κοινοί ε, κανόνες του ενοχικού δικαίου θα ε, από το δικαστήριο, από το ΔΕΚ. Αυτός ο δυνηρός και μακρύς δρόμος που αναφέρατε, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε σε δύο μήνες γιατί πραγματικά θα χρειάζονταν πολύ παραπάνω, πολλές παραπάνω διατάξεις στο κεφάλαιο αυτό. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχουν κάποιοι δικαστές οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτή τη δουλειά τελικά, σε τελική ναι. ανάλυση. Και αν δεν μπορούμε να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, ο καλύτερο δρόμο ποιο είναι η στοχοθετημένη εναρμόνιση. Mm. Έντονα στοχοθετημένη. Αυτή η εναρμόνιση και το είπε αυτό και ο κύριος Πέτρικ. Ε, θεωρώ ότι αποτελεί την ε, χειρότερη λύση και να δώσω κάποιες πληροφορίες παραπάνω, κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Εγώ είμαι Ευρωπαϊο νομικός και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει η εφαρμογή κοινών προτύπων χωρίς να εφαρμόζονται κοινοί κανόνες. Και είμαι σχεδόν βέβαιο ότι το ίδιο πρόβλημα θα είχαν και όλοι οι συναδελφοί μου και ότι το ΔΕΚ θα αντιμετώπιζε πολύ μεγάλα προβλήματα. Σας ρωτώ λοιπόν. Η γερμανική νομολογία για τις ε, τα επιτόκια μπορεί να διατηρηθεί. Θα μπορούσε να διατηρηθεί. Είναι πρότυπο το οποίο θα καταρακούσε το κεφάλαιο 4 ή όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε αυτό. Δεν είναι. Πιστεύω ότι πάντα το δίκαιο αυτό, η νομοθεσία αυτή καταρτίζεται ενάντια κάποιες κατάστασεις. Αυτό είναι κάτι κλασικά γερμανικό. Στην Αγγλία, και παράδειγμα, δεν, συμβαίνει. Χρειαζόμαστε λοιπόν τυποποιημένου όρους και θα μπορούσαν να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα και αν είναι διαφορετικά τα ήθη και τα έθιμα για να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος Σβάμπ. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήταν πολύ διαφορετικά τα έθιμα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το δίκαιο περί εκμισθώσεων. Ναι, μεν είναι δύσκολη αυτή η οδός, αλλά μπορούμε να την επιλέξουμε. Νομίζω ότι μία μέγιστη ενοποίηση και εναρμόνιση θα ήταν και δύσκολη στην κατανόηση από τους νομικούς και δύσκολη στην εφαρμογή και δεν βοηθά τον κανέναν τελικά. Είπατε ότι θέλετε να αυξηθεί η αξιολόγηση εξάντα των σημαντικών όρων, παρά να υπάρχουν τελικά ε, ε, εκ των υστέρων διαφωνίες. Στο νομικό μου σύστημα, οι πιο πολλοί όροι περνούν από τον δικαστικό μηχανισμό γιατί θα καταλήξουν τελικά στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Γερμανία, το οποίο θα πρέπει να αποφανθεί. Ο λόγος ποιος είναι, ότι οι εμπορευόμενοι καταρτίζουν τους όρους, τους συμβατικούς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα διατάξεις, αλλά όπου θεωρούν ότι υπάρχει κάποια ασάφεια. και κανένα ένομο μέσο δεν θα μπορούσε να τους βοηθήσει εκ των προτέρων. Θέλουν να ξέρουν τελικά τι θα αποφανθεί το δικαστήριο, γιατί ε, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν προ την ποιότητα των όρων. Θα πρέπει να εξετάσουν ποιο είναι ο χειρότερο όρο για του καταναλωτέ. Και η ίδια κατάσταση θα επικρατούσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε σχεδόν όλοι οι όροι τελικά να καταλήξουν ενώπιον του 10. Και αν το 10 δεν θα μπορούσε ούτε καν να εφαρμόσει ένα κοινό πρότυπο. Δεν θα μπορούσε να ε, επιβάλλει κοινού ε, κανόνες σε όλη την Ευρώπη. Θα είχαμε διαφωνίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να διευκολύνουν τελικά κανέναν. Και ιδιαίτερα οι εμπορευόμενοι δεν θα επέλεγαν το μοντέλο σας, γιατί δεν θα ήταν βέβαιοι για το κατά πόσο ένας συμβατικός όρος ε, είναι έγκυρος ή μη. Δεν θα κάνω και, και άλλα σχόλια, αλλά αν θέλετε, αν έχω πιο πολύ χρόνο, μπορώ να σας απαντήσω και σε άλλα ερωτήματα. Ε, αυτό θα μπορούσε να το πει ο καθένα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις αφέστατες σας παρουσιάσεις και για τον ενθουσιασμό με τον οποίο συμβάλλατε στη συζήτηση. Μπορεί να σας υποβληθούν στο μέλλον και γραπτά ερωτήματα και σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερως. Και τώρα κυρίες και κύριοι Σας άφησα να μιλήσετε γιατί είχαμε εδώ τους καθηγητάς, αλλά έχουμε και άλλες γνωμοδοτήσεις. Για να δω αν και δεν βλέπω. Πολύ ταιριαστό που θα μιλήσουμε για ρήτρες ηλιοβασιλέματος. Για την έκθεση Βάιλερ πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες που σε λίγο λίγη διορία τους. Μόλις έμαθα ότι υπάρχει μια πρόταση για smart regulation και στην πρόταση της Κομισιόν γίνεται και παραπομπή στην Επιτροπή μας ως προς την πρότασή μας να εξετάζουν συστηματικά οι συντονιστές τις αξιολογήσεις της Κομισιόν. Δεν την έχω εδώ βέβαια την επίσημη αυτή δήλωση, αλλά τέλος πάντων είναι ο κύριος Μπουζό εδώ με τη γνωμοδότησή του για την πολιτική ανταγωνισμού, αλλά η γραμματεία μου λέει ότι να αρχίσουμε μεν τη συζήτηση σήμερα, αλλά και στην επόμενη συνεδρίαση να τη συνεχίσουμε γιατί η διορία κατάθεσης τροπολογιών λίγη μετά την επόμενη μας συνεδρίαση. Κύριε Μπουζόη, συμφωνείτε, το δέχεστε, να αρχίσουμε απλώς σήμερα και να συνεχίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση, αφού θα είστε εκεί. Δεν θα είστε. Να αρχίσουμε με τη γνωμοδότησή μου. Όχι, όχι. Η κυρία Βάιλερ πρώτα είπα απλώς Συμφωνώ, συμφωνώ πρόεδρε, συμφωνώ. Μερικά λόγια τώρα και τα υπόλοιπα την επόμενη φορά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι και την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερο χρόνο αφού έχετε χρόνο για τις τροπολογίες. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία τότε. Λοιπόν, η κυρία Βάιλερ για τη γνωμοδότηση της... Ε, ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι το θέμα σας αφορά και προσωπικά. Προσωπικά. Κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι χαίρομαι για το γεγονός ότι δίνεται μεγάλη προσοχή στην έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι αμυγός τεχνικής φύσεως, ούτε είναι μόνο εσωτερικά, αν θέλετε, έχει εσωτερική σημασία για το, τη δική μας δουλειά. Επηρεάζει και την ε, δημόσια σφαίρα, το κοινό, το οποίο παρακολουθεί τις εργασίες μας. Είπατε δικαίως ότι η Επιτροπή μας είναι... επηρεάζεται ιδιαίτερα από το θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Και άκουσα αρκετά επικριτικά σχόλια και σε κάποιου τομείς ίσως και να ακούσαμε μάλλον ίσως και να είδαμε και θετικά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν οι προτάσεις μου δεν είναι και ιδιαίτερα επικριτική η πρότασή μου όσο θα περίμενε η Επιτροπή. Ωστόσο να πω ότι φυσικά και ισχύει αυτό που λένε και κάποιοι συνάδελφοι ότι παλαιότερα δεν ήταν ασυνήθιστο και είμαι προσεκτική εδώ να εκπονεί μελέτες αντικτύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την σταθεροποίηση, τη διασφάλιση, αν θέλετε, την πολιτική διασφάλιση των νομοθετικών προτάσεων της και να μην ελέγχει εναλλακτικέ λύσεις. Αλλά θεωρώ ότι αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν. Και εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί και όσα επιθυμούμε εμείς. Και το ελεγκτικό συνέδριο Θεωρεί ότι το σύστημα που εφαρμόζουμε είναι υποδειγματικό σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσως να είναι λίγο υπερβολικό αυτό, γιατί και οι Αμερικανοί κάνουν πολύ καλή δουλειά, ωστόσο να πω ότι κάνουμε πιο πολλούς ελέγχους αντικτύπου από ότι σε εθνικό επίπεδο, από ότι στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, γιατί ε, τα εθνικά κράτη κάνουν βασικά cost-benefit ανάλυση. Η Γερμανία θέλει τώρα να το επεκτείνει αυτό και να συμπεριλάβει και τις ε, επιπτώσεις στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και ούτω καθεξής, αλλά πάντα μιλάμε για οικονομική ανάλυση και μελέτη αντικτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέβαλε μια ανακοίνωση γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για τον πυλώνα της καλύτερης νομοθεσίας. Πολύ σημαντικό και ορθό αυτό. Ωστόσο, αναμένουμε να συμπεριληφθούν στη συζήτηση αυτή και κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία. Να κάνω λοιπόν κάποιες προτάσεις σε ό,τι αφορά και την δική μας Επιτροπή. Ως τώρα έχουμε την εντύπωση ότι οι ενώσει καταναλωτών και ότι οι επιπτώσεις ε, στην πολιτική για τον καταναλωτή δεν έχουν ληφθεί ακόμα επαρκώς υπόψη. Αυτό δεν ε, είναι δύσκολο να το αλλάξουμε και είμαι πεπισμένη ότι θα είναι δυνατόν να το πετύχουμε αυτό. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλεύεται συστηματικά με όλους τους εμπλεκομένους φορείς για να εξετάζονται όλες τις πτυχές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και το καθεξής. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι, και το βρίσκεται αυτό στο σημείο 4, η εκτίμηση επιπτώσεων αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο, ένα κείμενο εν εξελίξη, το οποίο θα συνιστά βήματα της νομοθετικής διαδικασίας, γιατί είδαμε ότι στα σημεία όπου υποβάλλουμε σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει με πολύ ευέλικτο τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει μελέτες αντικτύπου σε ό,τι αφορά επίσης ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες ε, γραμμές. Ε, το περιμένουμε αυτό εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια. Αλλά σκόπιμο θα ήταν να τις δούμε τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές, γιατί από ό,τι ξέρω στο Αμερικανικό Κογκρέσο υποβάλλονται και τροποποιούνται με κοινοβουλευτικό έλεγχο τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς αυτό. Όχι πως δεν εμπιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να επικρατεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Το ίδιο συμβαίνει και με το Κογκρέσο, να δούμε και ποια κριτήρια ισχύουν. Γιατί σε θέματα διαφάνεια έχουμε κάποια προβλήματα. Και τελευταίο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εξή. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω καταλήξει ακόμα και θα ήθελα να με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι. Ξέρω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνεται εξωτερική ανάθεση εντελώς ανεξάρτητη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ίδρυμα, σε μια μονάδα, μια υπηρεσία. Δεν θα ήθελα να πάμε τόσο μακριά, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε ήδη στην διάθεσή μας, να τα εξυγχρονίσουμε, προτού κάνουμε τέτοια εξωτερική ανάθεση. Το κάνουν βέβαια αυτό στην Αμερική, πολύ καλό, αλλά στην Αμερική χρησιμοποιούν 3.000 άτομα προσωπικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε ρεαλιστικά να συσταθεί μια τέτοια υπηρεσία. Να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ίσως κάποια συγκεκριμένα τμήματα του, της μελέτης που θα μπορούσαν να ανατίθενται σε κάποια εξωτερική υπηρεσία γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. Αν υπάρχει λοιπόν τέτοια εξωτερική ανάθεση, θα πρέπει φυσικά να υπάρχει ανάλογη ποιότητα, να υπάρχει έλεγχος ποιότητας, εννοείται. Αλλά και εμείς ως Κοινοβούλιο θα κάναμε τέτοια ανάθεση σε ιδρύματα, όπως για παράδειγμα τα ιδρύματα που εκπροσωπούνταν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανάλογα ιδρύματα θα, κατανε, θα ανέθετε την μελέτη δικτύπου αυτή. Άρα σε παράλληλη τροχιά θα κινούμασταν. Και αν τα αποτελέσματα ήταν ε, κακά, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει από συναδέλφους ότι δεν ε, ήταν θετικά, δεν ήταν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου, πολύ απλά δεν θα τους ε, ξαναχρησιμοποιήσουμε, δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουμε το εν λόγω ίδρυμα. Δεν ξέρω. Πριν από δύο εβδομάδε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είχε ταχθεί υπέρ τη εξωτερική ανάθεση. Αλλά υπάρχει και η άλλη εναλλακτική, να συμμετάσχουμε πιο έντονα και να δώσουμε σαφή εντολή στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, συμπερίληψη και την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή για καλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη διαφάνεια και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας. Αλλά δεν έχω ακόμα καταλήξει. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Ευχαριστώ. Very much indeed, uh, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βάιλερ. Έχουμε κάποιον σκιώδη εδώ, τον κύριο Βάκαμπ, τον κύριο Κρόιτσμαν και εγώ για την ομάδα μου. Και είναι εδώ και ο κύριος Μάξιμος Άγγελος από την Κομισιόν. Για να κάνουμε ένα γύρο λοιπόν σχολείων από τους σκιώδης. Πρώτο ο κύριος Βαντερκάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω λίγο στα Ολλανδικά. Γιατί είναι νομικά ε, σημαντικό το θέμα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους κατάλληλους όρους. Και εγώ διάβασα το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων και όντως μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι σημαντικά πιο επικριτική στη στάση της από ότι η κυρία Βάιλερ. Γνωρίζω όμως ε, την κυρία Βάιλερ. Μπορεί να προσθέσει σε ε, μετέπειτα χρονική στιγμή περαιτέρω κριτικά, επικριτικά στοιχεία. Ε, τρεις ερωτήσεις έχω. Κατά πρώτον, μπορούν οι μελέτες αντικτύπου να καθορίσουν την πολιτική, γιατί έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει απαραίτητα υπόψη τις μελέτες αντικτύπου. Είναι υποχρεωτικοί, δεσμευτικές αυτές οι μελέτες. Στα αγγλικά αναφέρεται η ανάγκη για μελέτες αντικτύπου. Μήπως θα έπρεπε να αναφέρεται η αναγκαιότητα για τη μελέτη αντικτύπου. Δεύτερη ερώτηση. Οι σύμβουλοι. Από ό,τι κατάλαβα, συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά αναθέτουν τις μελέτες στους ίδιους, ε, στα ίδια ιδρύματα. Αυτό μήπως θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε, δεν μπορεί να καταστεί φυσικά υποχρεωτικό, αλλά είναι κάπως περίεργο ότι και οι δύο χρησιμοποιούμε τους ίδιους συμβούλους. Ελπίζω να καταλήγουμε και στα ίδια αποτελέσματα. Τέλος, Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το outsourcing, Σύμφωνα με την κυρία Βάιλερ να το κοιτάξουμε αυτό με προσοχή γιατί με προβληματίζουν τα κοινοβούλια που κάνουν εξωτερική ανάθεση για τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό και θα ήθελα να υποστηρίξω τις ε, σκέψεις που εξέφρασα. Ευχαριστώ. Thank Van der Ευχαριστούμε κύριε Βαντερκάμπ. Κύριε Σκρότσμαν, ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Να πω καταρχάς ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον μία οδηγία, ένας κανονισμός θα βοηθούσε την ενιαία αγορά και αν δεν βοηθούσε να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει. Γιατί αλλιώς δημιουργείται ε, γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερο θέμα. Υπάρχουν νομικοί. Για παράδειγμα, υπάρχει στη Γερμανία νομοθεσία για την προστασία της μητέρας, για την προστασία των ε, γονικών δικαιωμάτων. Και φυσικά εξετάζουμε πώς θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάζει τέτοια θέματα σε ό,τι αφορά τυχές αναθέσεις συμβάσεων. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ καλό αν υπήρχε δυνατότητα έντονότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ή να προσθέσει κάποια στοιχεία του Κοινοβούλιο σε αυτά που θα έπρεπε να ερευνηθούν. Και πάντα θα έπρεπε να το εξετάσουμε αυτό από οπτική γωνία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί επειδή έχω εργαστεί σε μεγάλη επιχειρήση επί δεκαετίες και ξέρω ότι οι μεγάλε εταιρείε μπορούν να ανταπεξέλθουν χωρί κανένα πρόβλημα γιατί έχουν ειδικά τμήματα και σε πολλές περιπτώσεις οι μεγάλες εταιρείε ε, βοηθούν και τις μικρές ε, επιχειρήσεις που δεν έχουν τα μεγάλα νομικά τμήματα ή τα μεγάλα επιστημονικά τμήματα, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να εκτιμήσουν τις συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, στο σημείο 7 κυρία Βάιλερ, το γεγονός ότι αναφέρεστε ρητά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτό το γραφειοκρατικό άκτος θα τις επιβαρύνει. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η γραφειοκρατία να έχει να κάνει να εξαρτάται από τον αριθμό των απασχολούμενων. γιατί τις μεγάλες εταιρείες το γραφειοκρατικό άχθος αυτό είναι πολύ μικρότερο ανά υπάλληλο σε σχέση με τις μικρομεσαίες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημείο 7. Και φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε, κυρία Βάιλετ, τις επιπτώσεις των καταναλωτή, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και φυσικά ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις που θα κληθούν να φέρουν το βάρος και φυσικά σε, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αν θέλετε. Και πάλι, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται σε πλανητικότερη θέση σε σχέση με τις μικρές. Άρα, θα πρέπει πάντα να, κοιτάξουμε, να κοιτάμε ε, τι, σημαίνει, τι σημαίνει νομοθεσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Uh, thank you very much, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρότσμαν. Έχω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Αλλά ένα πρακτικό ζήτημα Φαντάζομαι είναι νωρί ακόμη για να το απαντήσει η κυρία Βάιλερ. Είχαμε και την έκθεση της πρωτοβουλίας της κυρίας Νίμπλερ που αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα, μια συγκεκριμένη πτυχή του θέματος και λάβαμε την ε, ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευφυή e νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι ότι ήδη γίνονται απερχιωμένες ε, κάποιες ε, παράγραφη της έκθεσης Νίμπλερ. Μήπως θα πρέπει να τις προσαρμόσει και η εξασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων είναι, παρά είναι περιορισμένο θέμα. Και η κυρία Νίμπλερ δεν μας έπεισε γι' αυτό, ούτε για την αναγκαιγγύηση τους. Πάντως, επανέρχομαι στο δικό μας θέμα και στην έκθεση η γνωμοδότηση της κυρίας Βάιλερ που είναι πολύ επίκαιρη και χρήσιμη αλλά φυσικά θα εμπλουτιστεί με τροπολογίες. Πάντως συγχαρητήρια κυρία Βάιλερ που επισημαίνεται με σαφήνεια ότι το έγγραφο αυτό μελέτης επιπτώσεων θα πρέπει να είναι δυναμικό και οι μελέτες επιπτώσεων δεν είναι ένα γραφειοκρατικό πρόσκομα. Είναι τμήμα μια διαδικασία που θα πρέπει να καταλήγει σε απτά αποτελέσματα. Και όλε οι πληροφορίε και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μια μελέτη εκτιμήσεων επιπτώσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται ω κάτι που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει το κοινοβούλιο ή το ευρύ Θα πρέπει αυτέ οι μελέτε να είναι τμήμα τη ε, συνηθισμένη διαδικασία για την ε, παρασκευή ποιοτικών ε, νομοθετικών προτάσεων. Και με τη διερεύνηση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων και την κρίση των, την ανάλυση των επιπτώσεών τους, μπορούμε να καταλήγουμε σε πιο ποιοτικέ νομοθετικές διατάξεις. Και όπως είπα και προηγουμένως, η παράταση αυτής της διαδικασίας και η επίκληση της πίεσης χρόνου για αποφυγή τέτοιων μέλετων επιπτώσεων, αυτό το επιχείρημα κατά τη γνώμη μου είναι ανεδαφικό. Γιατί μία πρόταση νομοθετική που δεν συνοδεύεται από μία λεπτομεριακή και εμπρόθεσμη μελέτη των επιπτώσεών της είναι εξ αρχής μία βάσιμη πρόταση νομοθετική. Επίση υπάρχει το θέμα της ανεξαρτησίας που θα πρέπει να το εξετάσουμε στο πλαίσιο τη όλη διαδικασία και όχι ως κάτι απομονωμένο. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στην ανακοίνωσή της για την ευθύνη νομοθεσία προσπαθεί να αναλύσει και να σχολιάσει τα επιχειρήματα για περισσότερη ανεξαρτησία. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον και κατά την εξέταση έκθεση Νίμπλερ. Πάντω η κυρία Βάιλερ πολύ σωστά χρησιμοποίησε τον όρο αντικειμενικά κριτήρια, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, μια διαβεβαίωση ότι η πάλι τη ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντικειμενική και δεν περιορίζονται στο να προσαρμόσουν την ανάλυση των, με, των επιπτώσεων στα, στις προτάσεις τους. Η δική μου, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει η εσωτερική διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να εγγυάται για την αντικειμενικότητα, γιατί η αντικειμενικότητα είναι το εχέγγυο για ποιοτικά αποτελέσματα. Αυτά. Πάντω η γνωμοδότηση τη κυρία Βάιλερ επαναλαμβάνουν πολύ αξιόλογη και θα είναι χρήσιμη και για την Νομική Επιτροπή. Φαντάζομαι θα ε, εμπλουτιστεί, πάντω η ήδη η βασική τη ε, κατεύθυνση είναι σωστή και ελπίζω να ληφθεί υπόψη δεόντως από την Νομική Επιτροπή. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντζελίνο για σύντομα σχόλια. Μετά θα ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και θα δώσουμε και το, στον κύριο Μπουζόη τη δυνατότητα να μας παρουσιάσει τη δική του έκθεση. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Αντζελίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που μόλις είπατε για την μελέτη αξιολόγησης και για την ανάγκη κομισιών να χορηγεί κάποια βάση εξέτασης των προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η έλλειψη αυτών των αξιολογήσεων δημιουργεί ακριβώς το πρόβλημα. Η γνωμοδότηση που έχουμε μπροστά μας τονίζει σχεδόν όλα τα σημεία που έθεσε την περασμένη Παρασκευή και η ανακοίνωση της Κομισιόν. Και ας τα σχολιάσω αρχίζοντας με το τελευταίο. Η πρόσκληση δηλαδή της Επιτροπής σας σε άλλες επιτροπές να κάνουν τις αξιολογήσεις στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας. Κάτι που για την Κομισιόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς και για το ελεγκτικό συνέδριο που καταλαβαίνει ότι η μελέτη αξιολόγησης δεν χρησιμοποιείται καμιά φορά από το Συμβούλιο ή από το Κοινοβούλιο στην αρχή της διαδικασίας όπου είναι και το σημαντικότερο σημείο για να γίνει μια αξιολόγηση της ποιότητας της νομοθεσίας. Έπειτα η έκθεση, η ονομοδότηση δηλαδή, θέτει, και μερικά από τα κυριότερα θέματα όπως είπα της ανακοίνωσης, δηλαδή τη διαβούλευση, ουσιοδέστατο θέμα, λόγος για τον οποίο επεκτείναμε και την, την περίοδο 8 εβδομάδων, τη δίμηνη περίοδο και όλα τα συστήματα διαβούλευσης το εξή θα χρήζουν βελτίωσης και με οργανώσεις, θα γίνεται διαβούλευση και με οργανώσεις των καταναλωτών και καταναλωτριών και με άλλους ενδιαφερόμενους. Τώρα για το ότι οι αξιολογήσει αυτές πρέπει να θεωρούνται ένα ζών έγγραφο και αυτό πολύ σημαντικό. Όπως γνωρίζετε τα τρία όργανα συμφώνησαν στη διαθεσμική συμφωνία ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ιδιαίτερα ανέλαβαν τη δέσμευση να αξιολογούν. Και στην τελευταία της ανακοίνωση η Κομισιόν άφησε ανοιχτή τη δυνατότητα συνεργασίας με τα δύο άλλα όργανα για να υπάρξει μια ευρύτερη ανάλυση των αξιολογήσεων που θα κάνουν που είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία της όλης διαδικασίας και το λέει και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος Βαρόσο στην πρότασή του, στην ανακοίνωσή του, έκανε και την πρόταση της ανάλυσης εξ post. Γιατί για μια καλή νομοθεσία πρέπει να γίνεται όχι μόνο αξιολόγηση των προτέρων αλλά και εκ των υστέρων για να δούμε αν η νομοθεσία έχει επιφέρει τα αποτελέσματα που προέβλεπε και με τον τρόπο με τον οποίο προβλεπόταν και να δούμε και αν χρειάζεται καμία βελτίωση όπως περαιτέρω μείωση των διοικη, του διοικητικού κόστους. Για τις επιπτώσεις επίσης η προσέγγιση των τριών πυλώνων της Κομισιόν έχει γίνει δεκτή και από το Ελεκτρικό Συνέδριο και έχουμε στόχο, σκοπεύουμε να κάνουμε περισσότερη αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων μεταξύ των οποίων βέβαια πρέπει να δούμε και επί των καταναλωτών και καταναλωτριών. Τέλος, για την αλληλεξάρτηση, για την αλληλοσύνδεση, η ανακοίνωση είναι ρητή και σαφής και δείχνει ποια ακριβώς είναι η θέση της Κομισιόν. Θεωρούμε ότι το υπάρχον σύστημα επιτρέπει να επιτευχθούν τα οι που έθεσε ο πρόεδρος Βαρόσο. Και με τη δημοσίευση της γραμματότησης ε, board προσπαθούμε να πετύχουμε όχι μόνο περισσότερη διαφάνεια αλλά και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αξιολόγηση. Με τον τρόπο. Και αν δεν απατώμε, έχω τελειώσει εδώ, εκτός από το εξή ότι η Κομισιόν είναι φυσικά διατεθειμένη να έρθει και άλλη φορά για να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες και να απαντήσει σε τυχόν απορίες. Το δεύτερο σημείο είναι πιο γενικό και ίσως θα πρέπει στο μέλλον να το συζητήσουν οι συντονιστές τώρα που έχουμε την πρόταση περί εφιούς νομοθεσίας επιτάπητος. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ για μια ανακεφαλαίωση, γιατί δεν μας μένει και πολλούς χρόνος. Θα ήθελα να θίξω και ένα σημείο κριτικής, να κάνω μια κριτική. Υπερασπιστήκατε το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπατε ότι κάνουμε κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά δεν μα αρκεί αυτό. Δεν μα αρκεί. Θα ήθελα να είχατε σχολιάσει κάποιες από τις απαιτήσει που θέτω ε, στην έκθεσή μου και είχα μία συζήτηση με Σουηδούς επιχειρηματίες και είπαν ότι θα ήθελαν οι μεγάλες αντικτύπου να εστιάζονται πιο πολύ σε θέματα ανταγωνιστικότητα. Και είπα ότι καλά και άγια όλα αυτά, αλλά δεν μα αρκούν. Πείτε μα λοιπόν, ποια είναι η θέση σα πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει πιο πολύ το Κοινοβούλιο, όχι τώρα, σήμερα, αλλά θα ήθελα να μου το πείτε αυτό. Φυσικά δεν είμαστε κατά των ανάλυσεων εκ των υστέρων, Post. Και θέλουμε φυσικά να γνωρίσουμε ποιες είναι οι συνέπειες της νομοθεσίας μας, αλλά καταρχάς χρειαζόμαστε μία σταθερή βάση, μια στερεά βάση για τις μελέτες αντικτύπου. Και να πω στον κύριο Φαντεκάμπ το εξή. Εμείς ε, εδώ στην Επιτροπή μας χρησιμοποιούμε τις μελέτες αντικτύπου. Μπορεί να με τις στηρούμε βέβαια και να αποφαινόμαστε τελικά ότι ως Κοινοβούλιο θα υποστηρίξουμε άλλη στάση. Γιατί παντού υπάρχουν επιστημονικές απόψεις. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει διαφάνεια, αλλά πλήρη, η πλήρης ε, ανεξαρτησία δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Μας έχουν προειδοποιήσει και οι Αμερικανοί, αλλά να μας πείτε ποιο ίδρυμα, ποιο πανεπιστήμιο, ποιος καθηγητής τελικά θα ήταν υπεύθυνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να ξεχάσουμε το ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια εντελώς ανεξάρτητη αρχή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much, uh, Σας ευχαριστούμε, κύριε Βάιλερ. Να ορίσουμε την 3η Νοεμβρίου ως διορία για τις, τρο... για τις τροπολογίες και ίσως στην επόμενη συνεδρίαση καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε. Εσύντομια... συντομία, Μήπω η κυρία Νίμπλερ στο μεταξύ τροποποιήσει του όρου αναφορά τη δική τη έκθεση μετά την πρόσφατη δημοσίευση τη ανακοίνωση περιεφίου νομοθεσία. για να εξετάσουμε και αυτή την πτυχή. Άλλωστε η κυρία Νίμπλερ γνωρίζει ποια είναι η δική μου θέση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπουσόη για μια εισαγωγική μόνο παρουσίαση της δικής του γνωμοδότησης, γιατί η πιο διεξοδική συζήτηση της γνωμοδότησής του θα γίνει στην επόμενη μας συνεδρίαση, στις 26 και 27 Οκτωβρίου δηλαδή, ανάλογα πότε σας βολεύει καλύτερα κύριε Μπουσόη. Ούτως ή άλλως αποσιάζουν και όλες και οι ηγητές, οπότε μόνο μία ακροθυγής παρουσίαση θα γίνει. Ξέρω αν έχουμε και πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, υπάρχει εκπρόσωπος, οπότε θα μπορούσε να πει δυο λόγια για τη γνωμοδότηση. Ούτω ή άλλω έχουμε το πολύ πέντε λεπτά μέχρι το πέρα συνεδρίαση. Λυπούμε που σα τριμώχνω έτσι κύριε Μπουσόη. Θα είμαι λακωνικό γιατί ξέρω ότι επίκειται και δεξίωση, αλλά δυστυχώ θα απουσιάσω από αυτήν γιατί έχουμε συνεδρίες και οδησηγητές για τα δομικά προϊόντα. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή είναι πολύ θετική και Κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να χειριστεί καλά την πολιτική ανταγωνισμού του 2009 στα πλαίσια της κρίσης, να αφήσει τα κράτη-μέλη με μεγαλύτερη ελαστικότητα να λάβουν μέτρα για να μετριάσουν τα αποτελέσματα της κρίσης και να μπορέσουν να δώσουν την ευκαιρία σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις πιστώσεις. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να αποφευθούν απαράδεκτες τρευλώσεις ανταγωνισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εκ του σύνεγγυς να παρακολουθήσει την εφαρμογή τέτοιων ασφαλιστικών δικλείδων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό μας ε, βασικό ζητούμενο, την προστασία του καταναλωτή, θέλουμε με σωστούς μηχανισμούς επανόρθωσης ή εναλλακτικέ λύσεις να αποζημιωθούν τα θύματα των παραβιάσεων της πολιτικής ανταγωνισμού. Mm-hmm. ό,τι αφορά τον φαρμακευτικό κλάδο, τη φαρμακοβιομηχανία, θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους φραγμούς εισόδου για τα γενώσιμα φάρμακα και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία θα ήταν χρήσιμο και για αυτή την περίπτωση αλλά και για άλλε και θα πρέπει να δώσουμε μάχη για να υλοποιηθεί επιτέλου ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Και για τον ενεργειακό τομέα πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευρύνει και τον ανταγωνισμό ώστε να διαμορφωθεί μια εσωτερική αγορά ενέργεια και να έρθουν τα εμπόδια για του νέου παρόχου υπηρεσιών ώστε να μπορούν εύκολα να διεισδύσουν στην αγορά. Αυτά και προσβλέπω στη συζήτηση με τους οικοδησηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη μας συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπουσό και ευχαριστώ θερμά για την πολύ καλή σας γνωμοδότηση που καλύπτει αυτά τα βασικά σημεία. Κύριε Μπρόμς, θα θέλετε να πείτε δύο λόγια για να κλείσουμε τη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν δέχεται αυτή τη σχέδιο γνωμοδότησης και σημειώνουμε την υποστήριξη του συντάκτη για τις, στις προσπάθειες της Κομισιόν να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση που ήταν βέβαια ο κύριος στόχος των προσπαθειών μας πέρυσι. Χωρίς να αγνοούμε τα υπόλοιπα. Θέλουμε να, δια, να ε, τον εισηγητή, θα, θα πραγματοποιηθούν συνθήκες ίσων όρων στον αγώνα αυτόν και ό,τι αποφασίσαμε έγινε λεπτομερός και απαιτήσαμε από τις τράπεζες να κάνουν και αναδιάρθρωση. Στην Επιτροπή Εικόνων την προηγούμενη εβδομάδα ο Επίτροπος Αλμούνια ανέφερε ότι θέλουμε στις αρχές του 12 να γίνουν όλα αυτά. Όσο για τη συνεργασία μεταξύ πολιτικής ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών και καταναλωτριών θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Κομισιό να δημιουργήσει ένα συνεπές νομοθετικό πλαίσιο και συνεργαζόμαστε στενά και με άλλες υπηρεσίες τη Επιτροπή, καθώς και με τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Βέβαια, πριν λήξει το φθινόπωρο θα τα τελειώσουμε όλα αυτά, δεν τα κάναμε